Good gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν βλέπω πολλούς ε, σήμερα. Δουλεύει το μικρόφωνο μου. Δεν βλέπω πολλούς βουλευτές εδώ, αλλά ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα σημεία στην ημερήσια διάταξη αύριο και σήμερα, αλλά να σας πω πρώτα κάποια πράγματα πριν ξεκινήσουμε. Καταρχάς, να σας θυμίσω ότι η συνάντηση μεταδίδεται στο web stream, όπως φαίνεται. Δεύτερον, να σας πω ότι τα πρακτικά της 27ης και 28ης Οκτωβρίου είναι διαθέσιμα, σας τα έχουμε στείλει. Ελπίζω ότι είστε σύμφωνοι, αλλά κάποιος θέλει να πει κάτι, κάποιο διαδικαστικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η ημερήσια διάταξη και έχω μια παρατήρηση για αυτήν να το πω γρήγορα. Στο σημείο 8 ένα έκτακτο ερώτημα στον, του Keith Taylor που δεν τον βλέπω πολύ συχνά εδώ και υπάρχει μια επαρκής απάντηση της, Κομισ... της Κομισιόν για αυτό το ερώτημα στα αρχεία μας Τέλος Οκτωβρίου είχε ήδη υποστείλει η Κομισιόν την απάντησή της. Γιατί λοιπόν τι θέλουμε εδώ. Ας βγει από την ημερήσια διάταξη. Και με εκπλήσει επίσης το σημείο 15. Είναι μια ομάδα από την ε, Γαλλία που θα μας επισκεφθεί. Εντάξει, αλλά μήπως στο σχεδιασμό να είμαστε λίγο πιο άμεσοι. Όταν έχουμε τέτοιες συναντήσεις με ομάδες όπως ας πούμε εδώ με το Παρίσι, ίσως θα πρέπει να το ξέρουμε εκ των προτέρων. Ναι, να έρχονται, αλλά αν η ημερήσια διάταξή μας είναι τόσο ασθενής που μπορούμε να την γεμίσουμε μόνο με τέτοια πράγματα, ας μην γίνεται τόσες μέρες η συνεδρία, ας γίνει μόνο μία μέρα. Προτείνω λοιπόν να βγάλουμε από τη ημερήσια διάταξη το σημείο 8. Κάποιο άλλο θέλει να μιλήσει αμέσω μετά, παρακαλώ. Δεν είμαι σίγουρος ότι αν συνήθως έχουμε 8, το σημείο 8 και τέτοια σημεία, αν τα έχουμε συνήθως στην ημερήσια διάταξη, ούτως ή άλλως θεωρώ ότι δεν είναι επαρκής η αλλως θεωρω οτι δεν ειναι επαρκή η απαντηση της Κομισιόν και είναι σημαντικό το θέμα στο Ενωμένο Βασίλε και θεωρώ ότι θα είναι και το κόστος μεγάλο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχει επανεγκατάσταση σε άλλα κράτη-μέλη και να υπάρχει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν όχι τόσο ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να είναι στη μερίσια διάταξη, αλλά ότι είναι ανεπαρκής η απάντηση της Κομισιόν και ίσως θα είναι μια ευκαιρία εδώ να δούμε τι ακριβώς έχει να πει η Κομισιόν. Να απαντήσω, Πρόεδρε. Πολύ σωστά λέτε, όμως ε, το θέμα είναι τι βάζουμε στην ημερήσια διάταξη. Κάποια πράγματα απαντώνται αμέσως. Γενικά δεν πρέπει να διωγγώνουμε την ημερήσια διάταξή μας με ερωτήματα των μελών. Συμφωνώ για το θέμα της επανεγκατάστασης που είπατε και ξέρω ότι και ο Πρόεδρος πραγματικά ενδιαφέρεται πολύ για αυτά τα θέματα, όμως ε, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αν γεμίζουμε τη μερίσια διάταξή μας με τέτοια ζητήματα. Το σημείο 8 λοιπόν όντως ε, είναι ατυχές που υπάρχει στη μερίσια διάταξη. Παρ' όλα αυτά, έχει δίκιο ο συνάδελφο ότι η γραπτή θέση της Κομισιόν εάν δίνονται χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επανεκατάσταση επιχειρήσεων, ε, είναι μη ικανοποιητική. Όπως και να έχει, θα πρέπει το θέμα αυτής της επανεκατάστασης να το εξετάσουμε πολύ στενά. Ναι, μεν έχει γίνει συζήτηση, υπάρχει ευαισθητοποίηση. Γι' αυτό παραμένει το σημείο 8 τουλάχιστον αν δεν έχετε αντίρρηση. Τώρα να συμφωνήσουμε και για το σημείο 15. Πραγματικά και εγώ εξεπλάγιν που είναι στην ημερήσια διάταξη, όμως έχουμε προς, προσκαλέσει τον κόσμο, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε έξω να περιμένει, αλλά την επόμενη φορά θα θέλω να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τη μερίσια διάταξη και πάμε στο σημείο 3, κάποιες ανακοινώσεις του Προέδρου. Από την κυρία Χιπνέρ. Όμως να πω ότι η συνάντηση των Υπουργών Μάλλον μόλις άκουσα ότι η κυρία Χιούμπνερ θα σας ενημερώσει όταν έρθει. Πάμε λοιπόν στο σημείο της ημερήσιας διάταξης 4. Ένα σημείο που έχει εντατικά προετοιμαστεί στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Ρωμά. Και εδώ, για αυτό το θέμα, καλό τον εισηγητή να παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να τονίσω και πάλι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη μειονότητα των Ρωμά στην Ευρώπη. Περίπου 12 εκατομμύρια Ρωμά στην Ευρώπη και οι περισσότεροι έχουν διαφορετικό τρόπο ζωή. Ένα μεγάλο αριθμό αυτή τη μειονότητα ζει υπό τη φτώχεια ή τη βαθιά ανέχεια και σε καταστάσεις κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού στην ε, ε, Ευρώπη οι πολιτικοί καταχρώνται την ε, θέση των Ρωμά για να πετύχουν κάποιους πολιτικούς στόχους. Ζούμε σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα, σε μια Ευρώπη ευημερία και είμαι πεπισμένο ότι δεν υπάρχουν μόνο εθνικές λύσεις πλέον. Αναμένω λοιπόν ότι τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ε, είναι συγχρονισμένα και θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση των Ρωμά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω συγκεκριμένε προτάσει προ αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα να ακούσω και σα ιδέε σήμερα. Α δούμε το χάρη το θέμα τη στέγαση. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκτηνε τι δυνατότητε παρέμβαση υπέρ ε, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων με ειδική αναφορά στου Ρωμά. Τα κράτη-μέλη μπορούν τώρα να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους και να χρησιμοποιήσουν έως το 2% του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη για το σκοπό αυτό. Όμως μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποίησαν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι λοιπόν τίθεται η ερώτηση γιατί το πράττουμε αυτό. Και αν τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν είναι πλήρω πεπισμένοι ότι είναι απαραίτητα αυτά μέτρα. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να συνοδεύσουμε τι προσπάθειε των εθνικών αρχών έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει αποτελεσματική συμπερίληψη των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Φυσικά πρέπει να γίνουν ε, κάποιε αξιολογήσει ε, στη στέγαση, πρέπει να βελτιώσουμε τι υποδομέ, τα συστήματα επικοινωνία κτλ προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί και ε, προκειμένου να μπορέσουν να μαθούν οι άνθρωποι να ψαρεύουν, παρά απλώ να του δώσουμε το ψάρι. Νομίζω ότι θα πρέπει τη στέγαση και τι άλλε κοινωνικέ παροχέ να τι συνδέσουμε με ε, την ε, εκπαίδευση των παιδιών και να δέχονται θέσει εργασία μέσω του θεσμού των διαμεσολαβητών. Αυτοί οι διαμεσολαβητέ για τι θέσει εργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό θεσμό για την καταπολέμηση τη ενεργία. Έχω λάβει επιστολές από τι οργανώσει του Ρωμά που ζητούν να μην συμπεριφερόμαστε πλέον στους Ρωμά σαν ευάλωτη κοινωνική ομάδα μόνο. Αναμένω μία μέρα να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα και ελπίζω στο εγγύ μέλλον. Αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να εγγυηθούμε την οικονομική και κοινωνική ένταξη, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στις θέσει εργασία και στι δημόσιε υπηρεσίε. Είμαι πεπισμένο ότι ε, και η περιορισμένη θετική διάκριση έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο. Κοινωνικός, ε, η κοινωνική αποδοχή των Ρωμά δεν είναι μόνο κοινωνική ευθύνη αλλά και οικονομική αναγκαιότητα. Δεν υπάρχει εναλλακτική πέρα από την πλήρη ένταξη των Ρωμά αυτό όχι ως πράξη φιλανθρωπίας αλλά προκειμένου ε, να εξυπηρετήσουμε τα οικονομικά συμφέροντα των χωρών όλοι και οι πολίτες και οι κυβερνήσεις ε, θα ωφεληθούν από ανθρώπους που έχουν καλύτερες δεξιότητες για να επιτελέσουν την εργασία τους. Ε, δηλαδή πρέπει όμως να έχουμε δύο κατευθύνσεις, πρέπει να υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές και από τη μειοψηφία και από την πλειοψηφία ε, η μελλοντική Ουγγρική Προεδρία ε, πρέπει να ασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 είναι απόλυτα σχετική πρέπει, καθώς επικεντρώνεται ε, στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην πρώιμη εγκατάλειψη του σχολείου. Η οικονομική κρίση εντείνει όχι μόνο τις δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τις διακρίσεις αλλά και τις δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την φτώχεια καθώς υπάρχει ανεπαρκής εκπαίδευση και λίγα προσόντα και το ο κοινωνικό αποκλεισμό. Θα πρέπει να στοχεύσουμε τα μέτρα μα στην εκπαίδευση και στη φοιτηση στο σχολείο, όχι μόνο ε, γιατί είναι λόγω τη εκπαίδευση, αλλά και επειδή κάθε χρόνο που περνάει ένα κορίτσι στο σχολείο σημαίνει ότι αναβάλει για ένα χρόνο το να γίνει μητέρα. Επίση, ε, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω τέτοια προγράμματα πέραν του 2013. Σήμερα περιμένω να ακούσω και προτάσει από εσά, αγαπητοί συνάδελφοι, για το πώ μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη συμπερίληψη των Ρωμά στην Ευρώπη. Και όπως ξέρετε, ε, υπήρξε και μία πρωτοβουλία, μία έκθεση πρωτοβουλίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ένταξη των Ρωμά και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση από την Κομισιόν και το Συμβούλιο για την νομοθετική πρόταση που αναμένεται το 2011. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Κόβατσετς. Πολύ ευαίσθητο το θέμα. Έχουμε μάθει ότι θα έχει καλύτερο, μεγαλύτερο δυναμικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει και καλό θα ήταν. Κύριο Φανιστέρο Ρόη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την άποψη που μας παρουσίασε. Είναι καλή η γνωμοδότηση, καλό το κείμενο και μένει στα πλαίσια της ε, περιφερειακής πολιτικής που γνωρίζουμε. Συμφωνώ με την προσέγγιση του. Θα ήθελα όμως να είμαστε λίγο πιο σκοπτικοί ως προς την Κομισιόν και τις εθνικές ε, κυβερνήσεις. Στο σημείο 4, για παράδειγμα, αυτό που λέει στο σημείο 4 του κειμένου σας. Όπως γνωρίζετε, στην αρχή του έτους Υιοθετήσαμε έναν κανονισμό για τους ευαίσθητους πληθυσμούς και με τους συναδέλφους θέσαμε μια σειρά ερωτημάτων πριν το καλοκαίρι Κάποια από αυτά απαντήθηκαν, αλλά όχι. Δεν ξαναμπήκαν στην ημερήσια διάταξη, όμως με βάση το περιεχόμενο αυτών των ε, απαντήσεων να πω ότι το πλαίσιο δείχνει ότι ως τώρα η Σύνοδος Κορυφής δεν έχει αλλάξει τα υφιστάμενα προγράμματα, όπως λέει το κείμενο. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί λοιπόν τα διαθέσιμα προγράμματα. 0,0%. Έτσι λοιπόν μέσα στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής η Κομισιόν θεώρησε ότι έπρεπε να παρουσιάσει μια σειρά πραγμάτων όπως τη χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Είμαστε στο τέλος του έτους. Συνειδητοποιούμε ότι το 2010-2011 θα είναι δύο χαμένα χρόνια. Και πραγματικά με ανησυχεί πολύ που δεν ασκούμε πίεση στα κράτη-μέλη και τις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν αυτά, αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτά τα κονδύλια. Η επίσκεψη της Επιτροπής ε, Περιφερειακών Υποθέσεων στην Ρουμανία, για παράδειγμα, δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες κοινότητες, ε, κάποιοι δήμαρχοι ε, που πραγματικά κάνουν πολύ σημαντική προσπάθεια για το σχολείο, την ε, στέγαση και την εργασία. Κάποια πράγματα αλλάζουν εκεί επί τόπου, όμως αυτό δεν είναι η γενική εικόνα. Γιατί λοιπόν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε τα κίνητρα στις υπόλοιπες πόλεις να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση. Ξέρω, για παράδειγμα, ότι υπάρχει στη Ρουμανία μεγάλη... Δεν χρησιμοποιούνται τα κονδύλια, μόνο 10% εξ αυτών χρησιμοποιούνται, άρα αυτό που γίνεται δεν είναι επαρκή. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί ε, στον τρόπο που προωθούμε την επικοινωνία μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που ζουν σε χώρες και σε πόλεις όπου μπορούμε να τους βοηθήσουμε θα πρέπει να βοηθούνται με τη χρήση των μέσων που είναι διαθέσιμα και αυτό δεν το έχουμε κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα είναι να γίνει μια προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιείται σωστά η συγχρηματοδότηση. Τουλάχιστον αν θεωρούμε ότι δεν ε, εξυπηρετεί σε τίποτα συγχρηματοδότηση, να έχουμε το θάρρος να το πούμε. Ευχαριστούμε. Κύριο κύριε ζητήσει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ καταρχήν τον εισηγητή για την ε, εργασία του. Είναι αλήθεια ότι η χώρα μου αντιμετώπισε το πρόβλημα προσφάτως και χαίρομαι που το ζητάνε τον Ρωμά αντιμετωπίζεται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας καθιστά αναγκαία ευρωπαϊκή παρέμβαση όσον αφορά τους νομάδες πληθυσμού. Εν γέννη. Καταρχήν χαίρομαι που το Περιφερειακό Ταμείο θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει σχέδια για την αποκατάσταση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, αν και όπως είπε ο κ. Βανίστηλ Ρόι, το κονδύλι αυτό υπάρχει αλλά δεν έχει εξαντληθεί. Δεν το χρησιμοποιούμε παρκώς. Θα έπρεπε να παροτρύνουμε τους Ρουμάνους συναδέλφους να κάνουν κάτι καλύτερο. Δεν είμαι υπέρ της ε, πολιτικής επωνομαδοποίηση, αν θέλετε, των ε, Ρωμά. Διότι ο ονοματικός χαρακτήρας είναι πολιτισμικό ίδιο χαρακτηριστικό αυτών των λαών. Οπότε δεν βλέπω γιατί, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, να αμφισβητήσουμε ακριβώ αυτό το ίδιο χαρακτηριστικό τους. Έστω και αν ορισμένα προγράμματα στέγασης έχουν ε, υλοποιηθεί σε διάφορες περιοχές. Επίση, το θέμα αυτό μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να ρυθμιστεί με σεβασμό τη αρχή τη ελεύθερη κυκλοφορία και με σεβασμό βεβαίω τη εθνική και κοινωνική νομοθεσία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ξέρουμε μια ισόρροπη λύση. Πέρα από τα στερεότυπα και τις υπερβόλες, γιατί ακούσαμε αρκετά τον τελευταίο καιρό, ε, είτε για τους Ρωμά, είτε για τις χώρες που του υποδέχθηκαν τη Γαλλία προκειμένου, για την οποία ε, το θέμα παραμένει εξαιρετικά λεπτό. Αυτά κύριε Πρόεδρε και κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάντσα έχει το λόγο. Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Να μην επαναλαμβάνω τόσα όσα ήδη υπόθηκαν. Σχετικά με τα όσα είπε ο συνάδελφος ε, Φανίστελ Ρόι, και εγώ θα πω, να χρησιμοποιήσουμε ακριβώ τους πόρους που είναι ήδη διαθέσιμοι. Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν χρησιμοποιούνται. Είναι κρίμα και είναι σοβαρό. Εξασφαλίζουμε σημαντικά ποσά, σημαντικά κονδύλια για τη στέγαση των Ρωμά, αλλά και για την εκπαίδευσή του, για τον πολιτισμό, για την απασχόληση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Συνεπώς, ας κινητοποιήσουμε τον μηχανισμό και παράλληλα ας δούμε γιατί υποχρησιμοποιούνται τα κονδύλια αυτά. Υπάρχει φαντάζομαι λύση. Μετά η ενημέρωση, η πληροφόρηση των Δήμων και των κοινοτήτων ή των οργανώσεων που εμπλέκονται σε τοπικό επίπεδο σε όλες τις χώρες. Στη Γαλλία, τη χώρα μου που γνωρίζω καλά, υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχουν όπως και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία τοπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν αυτούς τους πληθυσμούς. Χρειάζεται λοιπόν όλοι αυτοί οι εταίροι να ενημερωθούν καλύτερα, να τους πληροφορήσουμε ε, για τις δυνατότητες των Ευρωπαϊκών Ταμείων και να τους στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε. Τα κράτη-μέλη όμως έχουν και αυτά τον δικό τους ρόλο στην κινητοποίηση των ταμείων. Δυστυχώ δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, το ξέρω. και στι περιοχέ, στα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν ανοίξει αυτέ τι γραμμές του προπολισμού πρέπει να ενημερώσουμε του ενδιαφερόμενου ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά. Σήμερα δουλεύω πάνω σε μια έκθεση των στόχο 3. Λοιπόν υπάρχουν τα δύο περιφερειακά ταμεία. Α ενημερώσουμε, α δημιουργήσουμε του μηχανισμού ενημέρωση και να στείλουμε το μήνυμα, επαναλαμβάνω, ότι υπάρχουν κονδύλια τα οποία παραμένουν αχρησιμοποιητά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαντούλα έχει το λόγο. Πρόεδρε, να προσθέσω κι εγώ κάτι σε αυτήν τη συζήτηση στην Ρουμανία, αλλά όχι μόνο στη Ρουμανία. Η Ρέτζη, η επιτροπή μα στην Ρουμανία και δει στην δυτική Ρουμανία είδαν έργα υλοποιημένα υπέρ των Ρωμά. Θα άρχιζα όμω από ένα ερώτημα το οποίο δεν είχε απαντηθεί ούτε στην Ρουμανία ούτε αλλού. Γιατί δεν έχουμε μια εκτίμηση του συνολικού αριθμού των Ρωμά, γιατί οι διάφορε εκτιμήσει απέχουν εκατομμύρια ολόκληρα. Η δική μα εμπειρία στη δική Ρουμανία είναι εξή. Δεν έχουμε ακριβή εκτίμηση, γιατί οι Ρωμά θέλουν να ενταχθούν. Και οι Ρωμά, οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι, δεν δηλώνονται δεν δηλώνουν οι ίδιοι ότι είναι Ρωμά. Οπότε το ρήτημα επαναλαμβάνω, παραμένει. Γιατί δεν δηλώνουν σε αυτούς τους ως Ρωμά πλέον. Διότι θέλουν να είναι πλήρη μέλη της κοινότητας της χώρας στην οποία ζουν. Ταυτίζονται με το υπόλοιπο πληθυσμό του κράτους μέλους. Ας μην ξεχνούμε ότι στη Ρουμανία τουλάχιστον το 90% και περισσότερο των Ρωμά δεν είναι νομάδες. Έχουν εγκατασταθεί σε μόνιμες κατοικίες. Μόνο το 5, έστω ας πούμε 10% των παραμένουν νομάδες. Και βεβαίως δεν μπορούμε να τους ταυτίζουμε με εγκληματίε. Οι στατιστικές στην Ρουμανία δείχνουν ε, καταρχήν ότι οι Ρωμά εμπλέκονται στο μικρό έγκλημα σε... και όχι σε σοβαρά δεχθεί εγκλήματα ενδεχομένω. Η απάντηση για μένα και η λύση είναι εκπαίδευση, δουλειές και στέγαση. Όσον αφορά τώρα την ε, χρησιμοποίηση, την εξοποίηση των ταμείων, συμφωνώ πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο για την απορρόφηση αλλά και για την μείωση της γραφειοκρατίας για αυτούς που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τα σχετικά κονδύλια. Είχαμε έργο στη Δυτική Ρουμανία που δήμαρχος έκτισε πάνω από 280 σπίτια μένουν ήδη πάνω από χίλιοι Ρωμά. Και αυτό το κατόρθωσε με τοπικούς πόρους. Παραλαμβάνω πάνω από 280 σπίτια. Με χρήματα από τον προπολισμό του Δήμου. Και έτσι απέφυγε όλη τη γραφειοκρατία που συνεπάγεται προσφυγή σε κοινοτικά ταμεία. Είναι ένα δήμαρχο ο οποίο έχει μακρά εμπειρία βεβαίω σε κοινωτικά έργα, πρέπει να πω. Οπότε, Ας απλουστεύσουμε τις διαδικασίες προσφυγής στα ταμεία για τους Ρωμά. Αυτό είναι προτεραιότητα. Βεβαίως, οι έλεγχοι θα γίνουν, οι επαληθεύσεις ε, θα γίνουν. Αυτό είναι εκ των Τώρα όσον αφορά την ενσωμάτωση, την ένταξη των Ρωμά, τουλάχιστον στην περιοχή από την οποία προέρχομαι εγώ, ε, οι Ρωμά πρέπει να σα πω δεν έχουν πρόβλημα να βρουν δουλειά. Υπάρχουν πολυεθνικέ, στι οποίε ε, ήδη εργάζονται εκατοντάδε Ρωμά. Σε μια συγκεκριμένη εταιρεία από του 4.000 υπαλλήλου, πάνω από 700 είναι Ρωμά. Η εταιρεία αυτή έχει μάλιστα την πρόθεση να προσλάβει περισσότερου. Και κλείνω λέγοντα το εξή. Κατά την άποψή μου, ενσωμάτωση ένταξη σημαίνει και πάλι εκπαίδευση θέσεις εργασίας στέγαση. Και προς τούτο χρειάζεται φυσικά χρησιμοποίηση των κοινωνικών κονδυλίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε ματούλα. η κυρία Σμακοβά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το λόγο. Πριν ε, δύο μήνες ε, περίπου, η δική μας πολιτική ομάδα, πέντε μέλη από τη δική μας πολιτική ομάδα, οι σοσιαλιστές, ε, επισκεφτήκαν τη Σλοβακία. Είναι γνωστό ότι η Σλοβακία είναι μία από τις χώρες με το μεγαλύτερο πληθυσμό σε Ρωμά. Εγώ προερχόμαι από το Κόσιτσε, όπου έχουμε αυτή την περιβόητη περιφέρεια του Λούνικο που είναι συγκεντρωμένος ο πληθυσμός στο Ρωμά, αλλά έχουμε και πάρα πολλά χωριά στην Ανατολική Σλοβακία με υψηλή συγκέντρωση σε πληθυσμό Ρωμά. Επισκεφτήκαμε κάποια χωριά όπου τα τελευταία πέντε χρόνια έγινε μια προσπάθεια ένταξης στο Ρωμά στην κοινωνία και εδώ πρέπει να συμφωνήσω με τους συναδέλφους ότι η συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή άλλα ταμεία θα πρέπει να είναι αντικείμενο συντονισμού κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει ανάγκη να ασκηθεί πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση και στην τοπική αυτοδίκηση στους δημάρχους γιατί είναι επιβεβαιωμένο ότι εκεί όπου αναλαμβάνει δράση η τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχουν ε, λιγότερα προβλήματα. Επισκεφθήκαμε δήμους με 300 Ρωμά όπου οικοδόμησαν μέσα σε πέντε χρόνια ε, τα σπίτια τους ε, οι ίδιοι και μετά από πέντε χρόνια δείχνουν σαν καινούρια τα σπίτια, τα παιδιά φύτουν τακτικά στο σχολείο. Και επίσης ε, υπάρχουν και δραστηριότητε ε, για τα παιδιά Ρωμά το απόγευμα και οι κάτοικοι του χωριού δεν ε, αντιμετωπίζουν τον πληθυσμό των Ρωμά ως προβληματικό. Όμως έτσι έχουμε και άλλα χωριά όπου υπάρχουν και 3.000 Ρωμά. Και εκεί δεύτερη γυμνάσια πρέπει να ανοίξουν, να ε, ανοίγουν σε αυτά τα χωριά και πρέπει να προσφέρουν εκπαίδευση στα παιδιά Ρωμά ε, προκειμένου να έχουν ε, και κάποια βασικά προσόντα τεχνικής φύσης, παραδείγματος χάρη. Αυτό λοιπόν είναι δυνατό μόνο όταν τις αρμοδιότητες τις έχει η τοπική αυτοδίκηση, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας εμπειρία. Σας ευχαριστώ. Έχουμε άλλον έναν βουλευτή που θέλει να μιλήσει και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να αναφέρω ότι ε, όσον αφορά τις επιτυχή, τα επιτυχή παραδείγματα ενσωμάτωσης των Ρωμά, έχω και εγώ ένα παράδειγμα. Εμάς η εμπειρία μας έδειξε ότι είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε τα παιδιά των Ρωμά και στην προσχολική εκπαίδευση. Στα τσέχικα δεν έχει μετάφραση προς τα αγγλικά. Δεν υπάρχει μετάφραση. Υπάρχει καμπίνα τσέχικη. Άλλη μία φορά λειτουργεί η μετάφραση. Μια πολύ σημαντική πτυχή της ε, επιτυχής, επιτυχούς ενσωμάτωση στον Ρωμά είναι η συμπερίληψη των παιδιών του στην προσχολική εκπαίδευση. Εγώ είμαι ε, σε θέση να σας δείξω ένα παράδειγμα από το Όλμιτς, όπου εδώ και 10 χρόνια έχουμε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα για παιδιά στον υπηαγωγείο, όπου εκεί τους διδάσκουμε τσέχικα. γιατί πραγματικά το πρόβλημα είναι ότι δεν επαρκούν οι γνώσεις τους οι γλωσσικές όταν ε, έρχονται στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν τους φέρνει σε διαφορετική ε, θέση από ό,τι την υπόλοιπη ε, κοινωνία. Αν λοιπόν μπουν στην προσχολική εκπαίδευση τα παιδιά των Ρωμά, θα έχουν το κίνητρο και οι γονείς και πραγματικά μετά από αυτό το παράδειγμα βλέπουμε πως υπήρξαν παιδιά που τελείωσαν ε, και το δημοτικό, κάποιοι και το γυμνάσιο με μεγάλη επιτυχία. Γιατί δυστυχώς ένα από τα μεγάλα εμπόδια στη ζωή των Ρωμά είναι η έλλειψη εκπαίδευσης και εμείς ως ε, η πλειονότητα ε, θα πρέπει να καταργήσουμε αυτή τη διαφορά. Όταν καταφέρουν με την εκπαίδευση οι Ρωμά να τελειώσουν το δημοτικό ή το γυμνάσιο, βρίσκουν και δουλειά στην αγορά εργασίας. Και γι' αυτό ε, και στην Τσεχία δεν βρίσκουν πολύ Ρώμα δουλειά, γιατί δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταντσίλα έχει το λόγο. În primul rând, Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσέγγιση του. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους Ρωμά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Συνεχίζουν να είναι μία από τις πλέον ευάλωτες μειονότητες στην Ευρώπη βρίσκονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια και γι' αυτό πιστεύω ότι το πρόβλημά τους είναι και δικό μας πρόβλημα και πρέπει να προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε χρησιμοποιώντας κοινέ μεθόδους και κοινούς μηχανισμούς. Ε, φυσικά οι εθνικές κυβερνήσεις ε, φέρουν υψηλή ευθύνη στο να εφαρμόσουν τους κανόνες. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρε πολιτικές. Αν θέλουμε να έχουμε συστηματικό αντίκτυπο στο να μειώσουμε τις διαφορές μεταξύ των Ρωμά και του υπόλοιπου πληθυσμού σε όλους τους τομείς, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην παροχή στέγαση και φυσικά στην υγεία η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να αξιολογούν τις πολιτικές τους σχετικά με, τους ε, πληθυσμούς, ε, με τον πληθυσμό Ρωμά. Αν ε, η εφαρμογή των πολιτικών αυτών ήταν αποτελεσματική σε ορισμένα σημεία, εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα με τον πληθυσμό Ρωμά και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση, στη στέγαση και στην ένταξη αυτού του πληθυσμού. Ευχαριστώ. Η Kommission, ob ein Vertreter dort kurz das Wort ergreifen möchte. Dankeschön. Ευχαριστώ. Δίνω λοιπόν το λόγο και στην Κομισιόν. Προέρχομαι από τη ΓΑΜΑ Δελταπασχόλησης, από την ε, Διεύθυνση Τη ε, απασχόληση και υπάρχουν εδώ και συναδελφοί από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ρίτζιο και όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε εκπροσώπους από όλες τις πολιτικές για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος και η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει αλλά και οι Υπουργοί του Συμβουλίου ότι το θέμα της συμπερίληψης στο Ρωμά είναι κοινή ευθύνη των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αναλάβουν Έχουμε ε, δράση για να διασφαλίσουμε την ένταξη στο Ρωμά. Φυσικά ε, προέκυψε και στη ζήτηση αυτή ότι είναι τερογενής ο πληθυσμός στο Ρωμά. Μιλάμε για τους νομάδες, ε, τους Αθήγανους, ε, και άλλους πληθυσμούς σε ορισμένες περιοχές είναι πλήρως ενταγμένοι αλλά γενικά ξέρουμε ότι είναι από τις πλέον αποκλεισμένε και περιθωριοποιημένες μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των Ρωμά για πολλούς λόγους και ακόμη και, σε, και οι χώρες που προσπάθησαν να μετρήσουν τον ακριβή όγκο του πληθυσμού το Ρωμά ε, για κάποιους λόγους δεν τα καταφέραν γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να δηλώσουν τον εαυτό τους ό,τι αφορά την περιθωριοποίηση αυτό έχει τεράστιο προσωπικό κόστος αλλά έχει και κόστος για την κοινωνία και φυσικά η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι υπάρχει τεράστια οικονομική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν κατορθώσουμε να διασφαλίσουμε την ένταξη στο Ρωμά. Αυτό αναφέρεται και στην έκθεση του εισηγητή και τονίστηκε και σε μια προσφατή έκθεση της Παγκόσμια Τράπεζα, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 αξιολόγησε όλα τα διαθέσιμα μέσα που έχουν τα κρατημέλη για να υποστηρίξουν την ένταξη στο Ρωμά και ε, τα μέσα χρηματοδότησης ε, και τότε είχαμε κάποια συμπεράσματα από το Συμβούλιο ότι υπάρχουν τα σωστά εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά πρέπει να τα καταστήσουμε πιο αποτελεσματικά σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο ως προς τη λειτουργία τους και αυτό φυσικά έχει να κάνει ιδιαίτερα με τα διαρθρωτικά ταμεία για να βοηθήσουμε ε, του η τοπική αυτοδιοίκηση να χρησιμοποιήσει καλύτερα του πόρου. Ε, Πολλέ πρωτοβουλίε έχει λάβει Κομισιόν και ορισμένε εκδηλώσει πέρσι στην Ουγγαρία, φέτο στην Ρουμανία, του χρόνου στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία, φέτο τον Απρίλιο. Ε, ε, δημοσιεύσαμε μία ειδική ανακοίνωση πολιτικής για την ολοένταξη των Ρωμά και αναφερθήκαμε και στην ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι ε, υπάρχει νέα δυνατότητα για το Ευρωπαϊκό Τομείο την Περιφερειακή Ανάπτυξη για την υποστήριξη της στέγασης και για την υποστήριξη της απασχόλησης και της εκπαίδευση και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δύο αυτά μέσα. Όπως ξέρετε τώρα η Κομισιόν εξετάζει στενά τη χρήση των πόρων από τα κράτη-μέλη και από τα διαφορετικά ταμεία. Στείλαμε μια ερώτηση στα κράτη-μέλη και τώρα αναλύουμε τα αποτελέσματα και η Κομισιόν θα λάβει μια πρώτη έκθεση από την Task Force για τους Ρωμά αργότερα φέτος. Η Κομισιόν κατόπιν θα παρουσιάσει μια ανακοίνηση τον Απρίλιο του 2011 για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές στο Ρωμά και θέλουμε ε, φυσικά να ε, εντάξουμε, ε, να πετύχουμε εκεί τους στόχους της στρατηγικής 2020 για τη μείωση της στόχια, της καταπολέμησης της εγκατάλειψης του σχολείου, της απασχόλησης και θέλουμε να συμπεριλάβουμε τους Ρωμά στις εθνικές στρατηγικές μεταρρύθμισης και να ενεργοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Η Κομισιόν θα κάνει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις και σε αυτή την προγραμματική περίοδο και στις επόμενες Κάποιο συζητητή αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Progress και στο έργο αυτό για την καταπολέμηση τη στόχια και ε, τη δημιουργία θεσμών πρέπει να συνεχιστεί. Κοιτάξτε, σίγουρα η διεύθυνση για την ισότητα επίση θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και ευχαριστώ τον εισηγητή για την υποστήριξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω τον κύριο Κόβατσετς αν θέλει να προσθέσει ένα τελικό σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους και την Κομισιόν για την παρέμβαση και τις ε, εισηγήσεις τους. Ε, πραγματικά είναι ετερογενής ο πληθυσμός, δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για όλα. Αυτό που δεν με χαροποίησε πολύ είναι ότι άκουσα πως αν υπάρχει συγχρονισμός ε, και ίδιο επίπεδο κατανόησης μεταξύ των διαφόρων διαφερόμενων μερών, όπως ας πούμε οι κυβέρνησεις, οι ε, κομισιόν, το κοινοβούλιο κτλ. Ε, τα τελευταία 20 χρόνια ακούω πολλά για σχέδια δράσης, στρατηγικές, συμπερίληψη των Ρωμά και καλή πολιτική θέληση για την ενσωμάτωσή τους, ε, όμως λίγα είναι τα αποτελέσματα. Ελπίζω η νέα μας προσπάθεια για άλλη μια φορά να μην έχει τόσο μικρά, τόσο λίγα αποτελέσματα και να βρούμε ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να υποστηρίξουμε την ενσωμάτωση των Ρωμά. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και όχι γραφειοκράτες. Όπως είπε ο κύριος Ματούλα, χρειαζόμαστε απλοποίηση και την υποστηρίζω αυτήν την απλοποίηση στις ε, παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα ε, για τη στέγαση. Αν είχαμε στην αρχή τουλάχιστον 100% ε, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν καλό, θα πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι και μετά να πάμε στη συγχρηματοδότηση. Επίσης ευχαριστώ για τη συμβολή σας σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση. Ε, που προετοιμάζει τα παιδιά των Ρωμά να μπουν στο σχολείο μαζί με τα παιδιά της πλειοψηφίας ε, του υπόλοιπου πληθυσμού. Πραγματικά πρέπει ε, τα παιδιά των Ρωμά να μιλούν τη γλώσσα της πλειοψηφίας της χώρας τους και αυτό θα βοηθήσει την ενσωμάτωση γιατί θα υπάρχει συμβολή και από τις δύο πλευρές, και από την μειονότητα και από την πλειονότητα του, πληθυσμού. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συμβολή σας. Ε, δεν ε, τον τροχό. Ε, ξέρουμε ε, ότι το πρόβλημα είναι η στέγαση, η εκπαίδευση, η εργασία. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμόσουμε τις λύσεις, πώς θα βρούμε ε, τον τρόπο να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τον κοινό μας στόχο και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Αντρέη. Πραγματικά η ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα που έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία ήταν πολύ επικοδομητική. Βλέπουμε στις συζητήσεις εδώ στο σώμα ε, πόσο μεγάλη είναι η σημασία που δίνεται στο θέμα. Αυτό πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Υπάρχουν κάποιες παρεβολές στο μικρόφωνο της Προέδρου που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Λοιπόν, 8 ε, Δεκεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίας είναι η προθεσμία και θα ψηφίσουμε στην συνεδρίασή μας τον Γενάρη. Ευχαριστώ πολύ τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συναδέλφους. Περνάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Άλλη μια φορά, ανταλλαγή απόψεων με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, Μικέλ Λανταμπάσο, προστάμενο της Μονάδας Θεματικός Συντονισμός και Ενοτομίας, στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, ο οποίος ε, θα μας παρουσιάσει την ανακοίνωση της Επιτροπής η Συμβολή της Πολιτικής για τη Συνοχή σε μια έξυπνη ανάπτυξη που εγκρίθηκε από την Κομισιόν αρχές Οκτωβρίου. Ο Μικέλ Ανταμπάσο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μας ε, καλέσατε για αυτή την ανακοίνωση εδώ. Θα να παρουσιάσω αυτή την ανακοίνωση, θα σας παρουσιάσω εδώ τους κύριους στόχους της ανακοίνωσης και θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα δράσεων που χρηματοδοτούμε σήμερα. Καταρχήν θέλω να πω ότι αυτή η ανακοίνωση είναι σημαντική γιατί υπεγράφει από τέσσερις επιτρόπους, ε, τους ε, τέσσερις επιτρόπους που έχουν αρμοδιότητες στο θέμα της καινοτομίας ε, και ταυτόχρονα έχουν αρμοδιότητες και για τη θεματική πρωτοβουλία για την καινοτομία. Και αυτή η πολιτική παρουσιάζεται την ίδια στιγμή που αποφασίστηκε και η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Επίσης, ε, στέλνουμε το μήνυμα ότι υπάρχει σύγκληση και συμφωνία μεταξύ των επιτρόπων να ακολουθήσουν την ίδια κατεύθυνση σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα και επομένως υπάρχει πραγματική βούληση να υπάρξει συντονισμός και συνέργεια δράσεων στον τομέα αυτό. Πιστεύουμε ότι στην εν λόγω ανακοίνωση παρουσιάζουμε ότι η πολιτική μας ε, μπορεί να είναι και πρέπει να είναι στην καρδιά ε, της στρατηγικής για το 2020, η περιφερειακή προοπτική και η συμμετοχή των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης ε, είναι ουσιαστική για να πετύχουμε επιτόπου τους στόχους της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 και επομένως να βελτιώσουμε την διακυβέρνηση που στο παρελθόν μπορεί να έλειπε. Ε, από ορισμένα οράματα που είχαμε για την Ευρώπη, όπως τη στρατηγική της Λισαβόνας λόγου χάρη. Αυτή η ανακοίνωση επίσης στοχεύει στο να παράσχει πρακτική καθοδήγηση, εργαλεία, ιδέες για το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι με έναν ε, τρόπο αποτελεσματικό προ το κόστο από την πολιτική συνοχή, πώ θα περάσουν στον τομέα τη καινοτομία. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ κατευθυντήριε γραμμέ για τι διαχειριστικέ αρχέ, είτε είναι οι εθνικέ κυβερνήσει είτε η τοπική αυτοδιοίκηση, για το πώ θα χρησιμοποιήσουν του πόρου. Ο πρώτο στόχο αυτή τη ανακοίνωση επίση είναι να πουλήσει μέσα εισαγωγικά την ενία των ε, ειδικών, ε, των, στα έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. Ε, και αυτή η ανακοίνωση σε αυτές τις τρεις λέξεις επικεντρώνεται. Πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική συνοχή για την πρόθεση της καινοτομίας και να πετύχουμε όσο δυνατόν καλύτερους στόχους. Και τέλος, θα μπορούσε κάποιο να θεωρήσει αυτή την ανακοίνωση ως ένα μεγάλο βήμα ε, για την ε, ευθυγράμμιση των πόρων ε, που ε, χρησιμοποιούνται στον τομέα της ε, καινοτομία, Μιλάμε για διάφορου πόρου και που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδιαίτερα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η καινοτομία έχει αναγνωριστεί ε, ως ένα κύριο συστατικό οποιασδήποτε προσπάθειας για την οικονομική ανάπτυξη στις περιφέρειες των κρατών μελών. Και όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια έχουμε μία πρόσφατη έκθεση του ΟΣΑ που λέει ότι οι δημόσιες πολιτικές αναγνωρίζονται ως χρήσιμες στον τομέα αυτό για να αντιμετωπίσουμε την αποτυχία στην αγορά και να προωθήσουμε αποτελεσματικά την καινοτομία σε όλη την επικράτεια όχι μόνο σε ορισμένα σημεία ε, όπου έχουμε ανάπτυξη τεχνολογίας, αλλά σε όλη την επικράτεια. Θα σας δώσω κάποιες ιδέες τώρα για τους βασικούς στόχους της ανακοίνωσης ε, πριν να περάσουμε στους πιο πρακτικούς τρόπους ε, για το τι θα κάνουμε με αυτές τις στρατηγικές, τις έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης. Καταρχήν η ανακοίνωση στοχεύει στις συνθήκες πλαισίου που θα διαπραγματευτούν στα πλαίσια των επόμενων εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμιση την επόμενη φορά. Αυτή η ανακοίνωση επίση δεν κάνει λόγο για βασική έρευνα, αλλά μιλά για την κοινοτομία υπό την ευρία έννοια. Μιλάει για συστήματα, περιφερειακά συστήματα καινοτομία και μιλάει για συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ε, για τις εταιρικέ σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επίσης ε, ε, πηγαίνει και πέρα από την τεχνολογία αναφέρεται και σε νέους τρόπους οργάνωσης της παραγωγής για την κοινοτομία στις υπηρεσίες και τα Θα σας τα αναφέρω αυτά σε λίγο. Επομένως, η έννοια της αλληλεπίδρασης των ΣΔΙΤ ε, ή το τρίγωνο της γνώσης είναι πάρα πολύ ουσιαστικά στοιχεία, αποτελούν την καρδιά αυτής της ανακοίνωσης. Το σημαντικό που πρέπει να υπογραμμίσουμε ε, είναι να κατανοήσουμε γιατί αυτή η ανακοίνωση και γιατί τώρα. Αυτό γιατί για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή ε, αφιερώνει το 1 τέταρτο του προπολογισμού της στην πρόθεση της καινοτομία, δηλαδή σχεδόν 86 δισεκατομμύρια ευρώ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόθεση της καινοτομία. Και από αυτά τα 86 δισεκατομμύρια, τα 2 τρίτα του ποσού αυτού ε, είναι ένα ποσό που είναι στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα χορηγηθεί σε διάφορες ε, δράσεις. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η στιγμή να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να μπορέσουν ε, ε, να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι πόροι αυτοί. Και Τέλος, ένας βασικός στόχος της ανακοίνωσης είναι να αποβευθούν οι επικαλύψεις και ε, της μίμησης αν θέλετε. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα κέντρο βιοτεχνολογία σε κάθε περιφέρεια. Δεν θέλουμε να αντιγράφουμε εδώ προσεγγίσεις Silicon Valley σε κάθε περιφέρεια. Δεν ε, λέμε ότι έχουμε ένα μέγεθος που κάνει σε όλους. Ο καθένας πρέπει να βρει το δικό του τρόπο. Δεν δίνουμε συνταγές παρέχουμε μεθόδους και διαδικασίες, ε, έχουμε απόλυτο σεβασμό γιατί γνωρίζουμε ότι πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάσταση σε κάθε περιφέρεια προκειμένου να χαρακτεί μια διαφορετική στρατηγική για την προώθηση της καινοτομία σε κάθε περιφέρεια και γι' αυτό αναφέραμε εδώ κάτι, παραθέτουμε κάτι που ελέγχθη από ένα σύμβουλο της κυβέρνησης Ομπάμα με την ε, νέα ορμή που έχουν καυτεί για την πρόθεση της καινοτομία και των κλάστερ καινοτομία. Είπαν ότι η καινοτομία μπορεί να καλλιεργηθεί αλλά όχι να διαταχθεί ή να υπαγορευτεί. Είναι λοιπόν η καινοτομία βασικό ερώτημα εδώ είναι βασικό θέμα ε, κατά πολλούς τρόπους. Είναι σχετική για την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών μας. Η καινοτομία σχετίζεται άμεσα με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η απάντηση είναι ναι. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι η πολιτική συνοχή και η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική δεν αλλάζει τους στόχους της, δεν διαστρεβλώνει τους στόχου της, δηλαδή για να έχουμε τομεακού στόχου Όχι. Η καινοτομία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής ανάπτυξη, γιατί αποτελεί προτεραιότητα για τι εταιρείε μα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και πρέπει να... Αν δείτε τα πλέον ε, πρόσφατες πληροφορίες, θα δείτε ποια είναι ο συσχετισμός μεταξύ καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Μπορεί να ρωτήσετε τώρα, ε, πρώτα είναι το αυγό, πρώτα έκανε κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Κοιτάξτε, ε, υπάρχει εδώ μια σαφής ε, κατανόηση από τη βιβλιογραφία και ε, από την πείρα που έχουν όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις ότι η καινοτομία αποτελεί ουσιαστικό συστατικό για την οικονομική ανάπτυξη. Δεν θέλουμε μόνο να έχουμε δρόμους και άλλου τέτοιου είδους υποδομές στις πλέον ε, ευάλωτες περιοχές, αλλά χρειαζόμαστε και την καινοτομία. Και θα σας δείξω εδώ ένα χάρτη Βλέπετε εδώ πώς εξελίχθηκε η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική με πολύ μικρότερα κονδύλια στις αρχές του 90 αυτή η πολιτική αφιέρωνε το 4% μόνο των πόρων για την πρόθεση της καινοτομίας ενώ σήμερα έχουμε φτάσει στο 25% των 344 δισεκατομμυρίων. Έχουμε λοιπόν τεράστια αύξηση και με απόλυτου και με σχετικού όρου για την καινοτομία στα πλαίσια της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και μπορούμε εδώ να εξάγουμε πολλά συμπεράσματα αλλά τουλάχιστον ένα θα σας αναφέρω οι περιφέρειες και εθνικέ κυβερνήσεις και σας παρακαλώ να θυμάστε ότι πάνω από το ίμιση ε, των πόρων ε, του Ευρωπαϊκού για την Περιφερειακή Ανάπτυξη είναι στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων, χρειάζεται για να αναπτύξουν στρατηγικέ, νέα εργαλεία πολιτική και νέο σκεπτικό, προκειμένου να μπορέσουν να επενδύσουν σε αυτό το τομέα. Γιατί είναι δύσκολο ο τομέα αυτό. Δεν ε, μιλάμε εδώ για τη διάνοιξη δρόμων, ε, αλλά για τη διάνοιξη του νου. Δηλαδή μιλάμε εδώ για την προώθηση κάποιων άειλων στόχων. Αν δείτε εδώ την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη, ε, θα δείτε ότι η πολιτική μας ε, αρμόζει καλύτερα στα σημεία που είναι με το ε, πιο ανοιχτό πράσινο. Χρειάζονται περισσότερο εκεί καινοτομία γιατί θα πανώνται λιγότεροι πόροι. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από την μελέτη για την καινοτομία θα βρείτε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι μισές ευρωπαϊκές εταιρείες θεωρούνται καινοτόμε, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχουν, ε, έχουν εισαγάγει σημαντικές υπηρεσίες στην αγορά στα τελευταία τρία χρόνια και το ένα τρίτο εξ αυτών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το πράττουν αυτό με συνεργασία με άλλους, δηλαδή με πελάτες, με προμηθευτές, ακόμη και με ανταγωνιστές, αλλά και με πανεπιστήμια, κέντρα τεχνολογίας κτλ. Και ε, εν ώψη αυτή της πραγματικότητας και αυτής της πολυπλοκότητας πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσει ε, για δύσκολες ε, πολιτικές και εδώ πρέπει να βοηθήσουμε τις εθνικές και τις κυβερνήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης να τα πράξουν όλα αυτά. Τώρα να ολοκληρώσω την παρουσίαση τη ανακοίνωση με κάποιες συστάσεις που συμπεριλαμβάνονται εδώ και θα σα αναφέρω ορισμένα παραδείγματα. Καταρχήν, πρέπει να δημιουργήσουμε καλύτερες και μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ του προγραμμάτος, του προγράμματος πλαισίου και του προγράμματος του Ευρωπαϊκού για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και του προγράμματος για την καινοτομία στο θέμα της ε, καινοτομίας. Ε, θα πρέπει να δράσουμε με ένα συμπληρωματικό τρόπο. Ε, σίγουρα η έρευνα για την αριστεία είναι κάτι πολύ σημαντικό και υπάρχουν ε, σήμερα ε, στην Ευρώπη ε, σε 30 περιφερειές συγκεντρώνεται συγκεντρώνονται ικανότητε υψηλή τεχνολογία, αλλά πρέπει να το προωθήσουμε αυτό σε μια ανταγωνιστική και παγκόσμια κλίμακα. Αλλά επίση πρέπει να βοηθήσουμε και τι εταιρείε, τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει σε όλε τι περιφέρειε και μέσω τη καινοτομία εν τέλει, για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην παγκόσμια οικονομία και αυτό θα γίνει και μέσω της καινοτομία. Δεν είναι μόνο μέσω της περικοπής του κόστους. Θα έχουμε διαφορετική καινοτομία που θα βασίζεται στην προσαρμογή των γενικών τεχνολογιών και όχι μόνο ε, στην πρωτοπόρο έρευνα. Έτσι λοιπόν ε, εδώ μαζί ε, με το πρόγραμμα καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητα και μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη μπορούμε να κινηθούμε σε αυτό το τομέα. Πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην χρηματοοικονομική μηχανική, δηλαδή να έχουμε περισσότερα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, ε, περισσότερες εγγύησεις. Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική σήμερα βασίζεται σε επιχορηγήσεις σε μεγάλο βαθμό και αυτό μας λένε και εταιρείε ότι πρέπει να κινηθούμε περισσότερο προς ε, την κατεύθυνση της ε, χρηματοοικονομικής μηχανικής. Ε, οι εθνικές κυβερνήσεις, τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν πάρα πολύ λίγες δυνατότητες που προσφέρονται στον κανονισμό για τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Να έχουμε το ίντερνετ, έχουμε κάποια άλλα προγράμματα ε, Διεθνική συνεργασία, ακριβώς ε, για αυτό το σκοπό αλλά προσφέρονται πάρα πολλές ευκαιρίες ε, στον κανονισμό για την περιφερειακή συνεργασία και αυτό είναι απαραίτητο σε αυτόν τον τομέα αλλά υπάρχει υποχρησιμοποίηση. Επίσης, ε, πιέζουμε για δημόσιες προμηθείες για την πρόθεση της ε, καινοτομίας. Ε, λέμε επίσης στις περιφέρειες όταν καταρτίζετε τα σχέδιά σας για τον τομέα αυτό χρησιμοποιήστε συστήματα αξιολόγησης ομοτήμων, χρησιμοποιήστε διεθνείς εμπειρογνώμονες, σας διερευνήσουμε νέους τρόπους για να υποστηρίξουμε περίπου χάρη τις προσπάθειες του προγράμματος πλαισίου. Και ας ε, χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τις δυνατότητες ε, ανταλλαγής διδαγμάτων μεταξύ των περιφερειών και των χωρών στην Ευρώπη. Σε αυτή την ανακοίνωση, ε, προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι και πρακτικοί, είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από οποιαδήποτε εθνική και τοπική κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουν όταν σκεφτόμαστε για αυτές τις, όταν έχουμε και αυτέ τι έξυπνε στρατηγικέ για την εξειδίκευση. Σε αυτούς του τομεί ε, το η εφετηρία είναι τα κλάστερ, οι ομαδοποιήσει είναι γνωστά τα κλάστερ, ε, από τη βιβλιογραφία δεν ε, είναι ένας καινούριο όρος. Το καινούριο είναι οι συμβουλές πολιτικής που δίνονται. Λέγεται τώρα ότι θα πρέπει να βασίζονται στην αριστεία τα κλάστερ αυτά και θα πρέπει να ε, αναπτύσσουν μεγαλύτερη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο στη διαφάνεια που δεν μπορείτε να δείτε και δεν ξέρω γιατί. Αναφέρουμε πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό μέσω της πολιτικής μας. Αναφέρουμε μία σειρά παραδειγμάτων ε, κλάστερ σε διάφορες χώρες και επίσης ε, θα είδατε ότι έχουμε ε, εκπονήσει κάποιες κατευθυντήριες μεθοδολικές γραμμές για τη δημιουργία έξυπνων συστημάτων, για το πώς θα αναπτυχθούν τα κλάστερ. Εδώ εμπνευστήκαμε σε μεγάλο βαθμό από το έργο που έγινε από την ε, Ένωση των Κυβερνητών στις Ηνωμένε Πολιτείες και συνεργαστήκαμε με τους Αμερικανούς για να προωθήσουμε και αυτές τις έννοιες ε, στις δικές μας περιφέρειες. Ένας ε, από τους λόγους γιατί τα κλάστερ είναι σημαντικά. Το 40% των ε, υπαλλήλων μας στην μεταπληκτική βιομηχανία είναι συγκεντρωμένοι σε διάφορες περιφέρειες και φέτος είχαμε μια ομάδα υψηλού, μια ομάδα επίπεδου εμπειρογνωμόνων η οποία τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο προσανατολισμό προς την παγκόσμια οικονομία. Ένα δεύτερο πεδίο παρέμβαση είναι ένα περιβάλλον, ε, επιχειρηματικό περιβάλλον που να είναι φιλικό προς την καινοτομία. Εδώ μιλάμε για επιχειρηματικότητα και για startup. Ε, μιλάμε για την πρόωθηση της πνευματικής ιδιοκτησίας με τα κεφάλαια ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Πορτογαλία. Στα τελευταία έξι χρόνια έχουν ε, πενταπλασιαστεί, ξαπλασιαστεί τα διπλώματα βρεσιτεχνίας. Κάποια άλλα τώρα ζητήματα για να έχουμε αυτό το περιβάλλον για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις είναι μέσω της προσέγγισης ε, voucher. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ε, περιφερειακού τεχνολογικού σχεδίου στο Λίμπρο στην Ολλανδία που προωθήσαμε την δεκαετία του 90. Ήταν πολύ δημοφιλές τελευταία και ταξίδεψε σε πολλές άλλες ε, περιοχές και το ενδιαφέρον εδώ είναι αυτό που λέει ο ΣΑ σε αυτή την παράθεση που έχουμε εδώ, ότι δηλαδή οι πολιτικές θα πρέπει να είναι έξυπνος συνδυασμός της έρευνας και της πρόθεσης υψηλής τεχνολογίας, αλλά και της κατανόησης άλλων ε, τρόπων καινοτομίας. Και Όλα αυτά σχετίζονται πάρα πολύ με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν οι ίδιες την έρευνα. Δηλαδή αυτά τα voucher είναι η απάντηση. Ε, Επίση, ε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην χρηματοδοτική μηχανική. Έχουμε ένα παράδειγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο για το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, Μιλάμε για τα ε, συνεργασία, επιχειρηματική συνεργασία των πανεπιστημίων. Αυτό είναι κάτι απολύτω απαραίτητο. Δεν μιλάμε μόνο για τη διαβίου μάθηση, αλλά και για ε, τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα για πώς χρησιμοποιήθηκαν ε, οι πόροι. Έχουμε παραδείγματος χάρη της και καινοτομίας του πρίγκπα της Ουαλίας ε, και είχαμε παραδείγματος χάρη εκεί ε, υποστήριξη από τα τοπικά πανεπιστήμια. Δηλαδή βάζετε την ευφυΐα μέσα σε μια εταιρεία, ανοίγεστε ε, σε διεθνές επίπεδο και συνδέστε και με ένα πανεπιστήμιο. Επίσης, ε, εδώ στριφόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θέλουμε να τονίσουμε ε, πόσο σημαντικό ρόλο ε, παίζουν αυτά τα εκολαπτήρια. Δηλαδή, έχουμε 25 χρόνια εμπειρίας και λέμε στις ε, κυβερνήσεις ε, πόσο σημαντική είναι η καινοτομία και η πολιτιστική τομής, ε, παραδείγματος χάρη, στο πώς μπορούμε να προωθήσουμε την αξία μέσω του design και έχουμε παραδείγματα που χρηματοδοτούνται από αυτή την πολιτική σε διάφορες περιφέρειες που αποδεικνύουν αυτά που λέμε. Και τέλος, ε, μιλάμε για τη σημασία του ψηφιακού θεματολογίου, της χρησιμοποίησης ε, του διαδικτύου ως ε, μέσο για την προετοιμασία, για τη διάδοση μάλλον της γνώσης. Μπορεί η γνώση να ταξιδέψει πιο εύκολα από το ένα μέρος στο άλλο. Και βλέπετε εδώ τα διάφορα αριθμητικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα δεν ε, υπάρχει και πολύ μεγάλη απορρόφηση αυτή τη στιγμή των πόρων. Ε, έχουμε κάποια προγράμματα που καλύπτουν πολλές περιοχές και λέγονται fast tracks. Δηλαδή πώς μπορούν οι περιφερειές να μάθουν η μία από την άλλη και να δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους προκειμένου να εφαρμόσουν ε, στη δική τους περιφέρεια τις καλές ιδέες που μαθαίνουν από τους άλλους. Εμείς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε ε, και εδώ και το ψηφιακό θεματολόγιο είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για την ε, πρώτη ΣΔΙΤ στη Γαλλία ε, που είχαμε εκεί μια χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ενός βριζονικού δικτύου σε όλη την επικράτεια και στις περιφερειακές και αγροτικές περιοχές και στη Λιθουανία είχαμε ένα πρόγραμμα για την ένταξη στην πληροφορική. Και επίσης έχουμε τις δημόσιες προμήθειες που είναι ζωτική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί το 16% του ΕΠ στην Ευρώπη διοχετεύεται μέσω των δημοσίων προμηθειών. Μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των εταιριών με ένα καλό τρόπο για την πρόθεση της καινοτομία μέσω των δημοσίων προμηθειών. Όχι μόνο δηλαδή απλώς να δαπανούν τους πόρους μας. Και θέλω να αναφερθώ τέλος σε αυτή την ε, έξυπνη εξειδίκευση προωθούμε την έννοια αυτή, αυτή την ομπρέλα όπου εντάσσονται όλοι αυτοί οι τομείς παρέμβασης που ανέφερα γιατί αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα δύο σχολών σκέψης. Καταρχήν έχουμε την υψηλή ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία ε, αναθεωρεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και προέκυψε αυτή η έννοια ότι οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης είναι κάτι απαραίτητο, αποτελούν προϋπόθεση για τις εθνικές κυβερνήσεις και τις περιφερειακές κυβερνήσεις ε, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τους πόρους για την κοινοτομία γιατί θα αποφεύγονταν έτσι επικαλύψεις και καταστάσεις όπου μια περιφερεια έχει παραδείγματος χάρη 25, ε, έχει 25 ε, κλάστερ και άλλα 25 ανήκουν ε, στην, μάλλον υπόκειται στην εθνική κυβέρνηση και κανένα δεν συνεργάζεται με το άλλο. και μπορούμε εδώ να κάνουμε κάποιες επιλογές ε, γιατί ε, ε, βρισκόμαστε και σε μια περίοδο κρίσης και πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιούμε κατάλληλα τους πόρους για την πρόθεση της κοινοτομία. και εδώ έχουμε μια εξήγηση τι εννοούμε με αυτό. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θέλουμε να σας πούμε ότι δεύτερη σχολή σκέψης είναι τα συμπεράσματα της έκθεσης Φαμπρίτσιο Βάρκα ε, ο οποίος ε, είπε ότι η έξυπνη εξειδίκευση είναι ένας τρόπος να χρησιμοποιήσουμε την, ε, την πολιτική περιφερειακή ανάπτυξης με έναν τρόπο κατάλληλο για την πρόθεση της καινοτομία. και η καινοτομία είναι απαραίτητη για όλες τις περιοχές. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να πείσουμε τις εθνικές κυβερνήσεις και τις περιφερειακές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν την έννοια αυτή, δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν ε, τίποτα σε αυτό το τομέα ε, και αυτό είναι κάτι καινούριο. Η Κομισιόν απλώς θέλει να πει ότι αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσετε για το μέλλον. Αυτό είναι το στρατηγικό πλαίσιο στο εσωτερικό του οποίου θα πρέπει να λάβετε τις αποφάσεις πολιτικές και είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε. Και αυτό είναι ένα από τα πρακτικά συμπεράσματα αυτής της ανακοίνωσης Κομισιόν. Θα συστήσει μια πλατφόρμα για τις περιφέρειες, εργαζόμαστε από αυτού για να παράσχουμε συμβουλές και καθοδήγηση για το πώς ε, θα ε, τα αναπτύξουν όλα αυτά που αναφέραμε και να υπάρχει και αναθεώρηση σε σχέση με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στον τομέα. Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης ε, υπερβαίνουν αυτά που είχαμε το 90 ε, της στρατηγικής γιατί εδώ δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο διεθνές πλαίσιο στην ανάγκη θέσπισης προτεραιοτήτων στην ανάγκη να εστιάσουμε σε κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Εδώ δεν μιλάμε για το σχέδιο ε, επιδοτήσεων από το κέντρο, από τις Βρυξέλλες ή από οποιαδήποτε πρωτεύουσα, δηλαδή να πούμε διαλέγουμε τους νικητές. Το αντίθετο ε, πρόκειται για μια διαδικασία που θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε επιχειρηματική ανακάλυψη. Δηλαδή πώς μπορούμε μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις και την τοπική να δούμε που ε, μπορούμε να επενδύσουμε για να προωθήσουμε καλύτερα την καινοτομία. Σας ευχαριστώ. like ευχαριστώ. Ξεκινάμε την συζήτηση. Μάρκος πίπε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και κύριε Λάμπερτ για την πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση. Θα ήθελα να μην ρίξουμε πολύ νερό στο κρασί μας, αλλά να θέσω κάποια ζητήματα. Έχουμε εδώ στην περιπτωκή, επιτροπή μας ε, θέσει κάποιους στόχους, ε, ε, τον στόχο 1, τον στόχο 2 που είναι πιο οριζόντιος και τον στόχο 3 που είναι πέρα από τα σύνορα. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ και δύο-τρία χρόνια είχαμε ενδιάμεσα αποτελέσματα που ήταν ε, έδειξαν μεγάλη επιτυχία σχετικά με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής ε, στις περιφέρειες αλλά και σχετικά με τις ανάγκες των περιφερειών. Είναι επιτυχημένη η πολιτική λοιπόν. Μιλάμε για το έξυπνο, την ε, έξυπνη ανάπτυξη, την αηφόρα ανάπτυξη, πρωτοβουλίες της στρατηγικής 2020 και θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω γιατί τώρα αλλάζουμε πλήρως ε, ρότα γιατί δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά που είναι οι ανάγκες των περιφερειών. Ε, οι περιφέρειες έχουν ανάγκες. Μιλάμε για εμπειρογνώμονες από οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Πορτογαλία. Όλα αυτά είναι καλά. Όμως, πού ε, βλέπουμε όμως αν αυτά ε, ας πούμε αντιστοιχούν στις ανάγκες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας κτλ. Όταν ε, δούμε τις επιπτώσεις αυτών που μας παρουσιάσατε, αν δούμε τι θα γίνει με το smart growth στο μέλλον και ε, ποιες είναι οι επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με αυτές τις διάφορες μορφές ανάπτυξης, οι οποίες είναι διαφορετικές, ε, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει από τη μία μια κεντρική διάθεση, μια κεντρική τάση και από την άλλη ε, οι περιφέρειες δεν ε, έχουν την ευκαιρία να γίνει ακουστός ο λόγος τους. Θα πρέπει λοιπόν εμείς ως Περιφερειακή Επιτροπή, Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων και Επιφερειακής Ανάπτυξης να διασφαλίσουμε ώστε αυτό να γίνεται. Ε, λυπάμαι, αλλά αυτή ήταν η εντύπωση που τουλάχιστον εγώ είχα από όσα μας παρουσιάστηκαν. Άρα Κομισιόν πρέπει να αποδείξει ότι είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από τη βάση. Ο κ. Φανίστελ Ρόι. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Μπορείτε να μας στείλετε και το κείμενο γιατί θα άξει να ξαναδιαβάσουμε τα όσα μας είπατε. Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 περιμένουμε ο καθένας, τα κρατημέλη και οι άλλοι να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια. Όμως, αυτά πρέπει να γίνουν με τη χρήση όλων των τεχνολογιών, των ευφυών τεχνολογιών, των πράσινων τεχνολογιών και ούτω καθεξής. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι πρώτο. Ποια θα είναι αιτία και ποιο το αποτέλεσμα. Τώρα αυτό για τον εξή λόγο. Πρώτον, έχουμε μια περιφερειακή διάσταση, η οποία προστέθηκε στη συνθήκη. Υπάρχει σχετική πράσινη βίβλος. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό τώρα είναι clustering ή συνεργατικό σχηματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Η κέντρα αριστείας. Εν πάση περιπτώσει αυτά όλα καλά είναι. Χρειάζεται σίγουρα η συνεργασία, ο συντονισμός και η επικοινωνία. Στα αγγλικά είναι τα τρία C. Και φυσικά χρειαζόμαστε και τις φυσικές υποδομές. Όλα αυτά παραλαμβάνουν πολύ ωραία. Όμως, βλέπω τώρα να εξειδικεύουμε την προσέγγιση μας προς της ευφυής όπως λέμε, τεχνολογίες. Και όλοι τρέχουμε προς τα εκεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε συνεχώς πολλές πρωτοβουλίες, δημοσίευσε ένα σωρό εκθέσεις, ιδιαίτερα στην Επιτροπή μας, για να εξηγήσει πώς βλέπει τα πράγματα. Εγώ λοιπόν θα σας παρακαλούσα να λάβετε λίγο περισσότερο υπόψη σας τη γνώμη του Κοινοβουλίου, διότι είναι σαν είμαστε όλοι πάνω σε ένα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος πηγαίνει προς μία μόνο κατεύθυνση, χωρίς, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τις άλλες παραμέτρους, την ίδια την περιφερειακή πολιτική. Προσπαθείτε νομίζω να βραχυκλώσετε την ε, διαδικασία. Εάν κινηθούμε υπερβολικά γρήγορα, φοβούμε ότι οι διαπραγματεύσεις με τα κρατή-μέλη, με τις περιφέρειες και με την Κομισιόν θα οδηγηθούν σε ένα διέξοδο. Κανείς δεν θα καταλαβαίνει τι γίνεται και ποιο κάνει τι. Επί της ουσίας, ναι, αν θέλετε μπορώ να συμφωνήσω. Είχαμε και την έκθεση του συναδελφού Κράτσεφ στην οποία υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα πράγματα. Όμως, η αρχιτεκτονική της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να λάβει υπόψη της τις πραγματικές δυνατότητες υλοποίησης. Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως, ε, αν μπορούμε να έχουμε το κείμενο να το ξαναδιαβάσουμε. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με όλα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Μάνα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάσο. Δύο πράγματα για την καινοτομία. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο τι ακολουθεί την καινοτομία. Γιατί η καινοτομία αυτή καθ' αυτή ως αυτοσκοπός δεν αρκεί. Πώς θα επωφεληθούμε από την καινοτομία, πώς θα υλοποιήσουμε εμπορικέ εφαρμογέ, πώς θα ανταγωνιστούμε τις ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα. Γιατί η προσπάθεια είναι μεγάλη κλίμακα στην Ευρώπη, αλλά θα είναι και τα αποτελέσματα αντίστοιχη κλίμακα με τι ΗΠΑ. χρειάζεται και σχετική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση αυτή πρέπει να είναι τμήμα της γενικότερης συζήτησης για την περιφερειακή πολιτική, την συνοχή και την καινοτομία βεβαίως. Αλλιώς φοβούμαι ότι τα ωφελήματα δεν θα είναι αξιοποιήσιμα. Γιατί αν κάνουμε και στην περιφερειακή πολιτική ότι κάναμε στην ε, Γεωργία, ίσως κάτι καλό να προκύψει. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε ένα πολιτές πλαίσιο και εν ώψη της ε, στρατηγικής του 2020. Να λάβουμε υπόψη μας ε, τις δημορφίες, τα χαρακτηριστικά των περιφερειών, τα ισχυρά του σημεία. Χάρη την συνοχή προχωρήσαμε με την ε, βιοενέργεια και την κοινοτομία σε διάφορες περιφέρειες. Μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι η ΣΥΤ είναι εξαιρετικά χρήσιμη, κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Ο συνάδελφος ε, έθεσε ερωτήματα που χρήζουν πάντως απαντήσεως και ελπίζω ότι θα βρούμε τέτοιου απαντήσει. απαντήσεις. Ευχαριστώ για την παρουσίαση καταρχήν. Γενικώ, η φιλοσοφία που διέπει αυτήν την παρουσίαση και την πολιτική του 2020 είναι λογικά πράγματα. Τώρα, αυτό που είπε ο Λάμπερτ ε, είναι σωστά. Πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες και στους άλλους εμπλεκόμενους ότι αυτά είναι ζωτική σημασία. Διότι αν δεν τα ενστερνιστούν αυτά οι πολίτες μας, δεν θα σημειώσουν πρόοδο. Δεύτερον, με βάση ποια κριτήρια αξιολογείται την καινοτομία και τα αποτελέσματά της συμβολή στο ΑΕΠ, νέες θέσεις εργασίας, νέα προϊόντα. Πώς μετράτε λοιπόν την πρόοδο. Και δεύτερον, μάλλον τρίτον, από 4% πριν από 20 χρόνια Έχουμε φτάσει στο 25% σήμερα στον τομέα. Και μας είπατε ότι ένα μεγάλο τομέα των κονδυλίων αυτών είναι στα χέρια των εθνικών και των περιφερικών των, των κυβερνήσεων και των περιφερικών αρχών. Πώς γίνεται αυτό, για εξηγήστε μας. Και τώρα η συνεργατική συμμετοχή είναι πολύ σημαντική. Τα στο Μανχάιμ που είναι μια σχετική μερίδα και Σαφώ η ανταλλαγή πληροφοριών, η μεταφορά γνώσης είναι πολύ σημαντική. Σίγουρα μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτού, οι οποίοι καινοτομούν ο καθένα στην περιοχή του. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τι γίνεται στι άλλε περιφέρειες. Συμφωνώ με την ιδέα. Η συνεργασία μεταξύ περιφερειών λοιπόν είναι πολύ σημαντική, διότι ακόμα και οι συνεργατικοί σχηματισμοί εντό συγκεκριμένων περιφερειών πολλέ φορέ ε, ζουν σε ένα στεγανό. Οπότε ένα λόγο παραπάνω. Είναι μάλιστα θα έλεγα ζωτική σημασία να έρθω σε επαφή με άλλε περιφέρειε. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά εδώ και όπω ζήτησε και ο Λάμπερ θέλω και εγώ την παρουσίαση γραπτό, γιατί έγινε πολύ γρήγορα και δεν θέλω να χάσω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πρόεδρος, ε, μας έστειλαν ήδη, την έχουμε την παρουσίαση αυτή, την παρουσίαση του κυρίου Λαντομπάσου, θα τη στείλουμε σε όλους και με την ευκαιρία να θυμίσω ότι είναι τμήμα της ανακοίνωσης της Κομισιόν που παρουσιάστηκε αρχές Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Είναι στα συνημένα της ανακοίνωσης. Υπάρχει το κείμενο δηλαδή, μην έχετε εμφολία. Και σας θυμίζω ότι και τον περασμένο μήνα συζητήσαμε και πάλι θέματα καινοτομίας στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Ο περιφέρεια της Νοτιοδυτικής Ολλανδίας ήρθε εδώ και μας μίλησε για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων για τους σκοπούς της καινοτομίας στο επίπεδο των περιφερειών. Και ακούσαμε για το φαινόμενο αυτό, δηλαδή σε πολλές περιφέρειες να ευνοούνται τα σχέδια καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε μια γενικότερη τάση λοιπόν υπέρ τη καινοτομία και προ την καινοτομία και μαθαίνουμε από όσου έχουν υλοποιήσει τέτοια έργα ήδη. Κύριος Αγκουράκης. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε απόλυτα δίκιο όταν λέτε ότι στην Επιτροπή μας ε, έχουμε όντως συζητήσει ορισμένες φορές, αρκετές φορές το ζήτημα αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματικά απασχολούμαστε με τέτοιου είδους ζητήματα. Καταρχήν θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να σε επαναλάβω αυτό που έχω πει και άλλη φορά, ότι εγώ δεν συμφωνώ η πολιτική της συνοχής να υποτάσσεται σε άλλους σκοπούς. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ δηλαδή σε αυτό που συζητάμε σήμερα, η συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή σε μια έξυπνη ανάπτυξη. Αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί εμάς και μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Λαμπαντάσου δεν το θεώρησε καν αναγκαίο να μας το πει, είναι πώς η έξυπνη ανάπτυξη θα συμβάλλει στην πολιτική συνοχής. Εμείς είμαστε μια, μια επιτροπή που ενδιαφέρεται να υπάρχει συνοχή σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από ό,τι γνωρίζω, κυρία Πρόεδρε, και νομίζω το ξέρουμε όλοι αυτό, όταν μιλάμε για καινοτομία, αυτό μας ενδιαφέρει είναι πραγματικά το τελικό προϊόν. Μια συνάδελφος το είπε πριν. Μας ενδιαφέρει τι ακολουθεί μετά την καινοτομία. Μας ενδιαφέρει το προϊόν. Αυτό, οι συνθήκες οι σημερινές λοιπά είναι τέτοιες που όλοι γνωρίζουμε και το μεγάλο κόστος για έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και όλοι γνωρίζουμε ότι για να είναι αποτελεσματικό το προϊόν χρειάζονται οικονομίες κλίμακας όπως ονομάζονται. Άρα οι περιφέρειες, αναρωτιέμαι ποιες περιφέρειες θα υπάρχουν μερικέ, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των περιφερειών δεν είναι καν σε θέση να δημιουργούν οικονομίε κλίμακα για τα προϊόντα που πιθανόν να προκύψουν από τι καινοτομίε του. Και δυστυχώ, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να σα πω, και το ξέρετε και εσεί νομίζω, ότι ο δείκτη ευρεσιτεχνιών δεν λέει και πολλά, πράγματα. Πράγματι, η Πορτογαλία ε, έχει εξαπλασιάσει τι ευρεσιτεχνίε τη. Και η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο αριθμό αλλά και οι δύο χώρες όπως ξέρετε είναι σε μια ε, πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση και αν θέλετε ακόμα και σε ζητήματα ανταγωνισμού όπως λέτε. Κατά συνέπεια υπάρχει ένα ζήτημα εδώ το οποίο δεν ξεκαθαρίζεται. Ένα δεύτερο ζήτημα που ανησυχεί πάρα πολύ είναι αυτό που άκουσα και φαντάζομαι ότι έτσι είναι, αλλά αναρωτιέμαι πώς θα γίνει αυτό. Μας είπε ο εισηγητής ότι είναι ανάγκη να καθοριστούν στρατηγικές προτεραιότητες για την καινοτομία στις περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναρωτιέμαι ποιος θα τις καθορίσει αυτές τις στρατηγικές προτεραιότητες, ποιος θα τις ελέγξει και με ποιες διαδικασίες θα αποφεχτούν αυτό που υπόθηκε να μην υπάρχουν υπερκαλύψεις. Τρίτο ζήτημα και πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που γίνεται λόγος για εξοικονόμηση πόρων, αυτό που με, με κάνει να απορώ πάρα πολύ είναι γιατί δεν γίνεται καμία αναφορά στο αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα ή κάποια κριτική μεταξύ συντονισμού ή όχι των προγραμμάτων καινοτομία σε επίπεδο περιφέρεια, αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμή, και του προγράμματο πλαίσιου για την έρευνα και ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μεγάλα τα ποσά εκεί. Γιατί δηλαδή να μην δει κανένα πώ μπορεί να εξειδικευθεί το πρόγραμμα πλαίσιο σε επίπεδο περιοχή, περιφέρεια αν θέλετε, και όχι να πηγαίνουμε τώρα από το μηδέν, όπου η τάδε επιχείρηση έχει ένα project, πάει σε μια τράπεζα, παίρνει ένα risk capital και τελειώνει, κυρία Πρόεδρε, γιατί βλέπω ότι ε, σας κουράζω. Ε, τελειώνω λέγοντας το εξής, ότι είναι ανάγκη κατά τη γνώμη μου να δούμε τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν. Είχα την τύχη της προάλλες να συναντηθώ με τους ε, συνδικαλιστές της Αλκατέλα από τη Γαλλία και μου είπανε κάτι, το ξέρουμε όλοι, δεν ανάγκη να σας το πω εγώ, ότι λόγω του ανταγωνισμού και αυτής της οικονομίας αγορά αγοράς και της παγκοσμιοποίησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον στον πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο των τηλεπικοινωνιών πλημμυρίζονται κινέζικα προϊόντα και ρωτάω, στο ζήτημα αυτό θα υπάρχει κάτι, χρειάζεται να δούνε και οι περιφέρειες τι θα κάνουν, διότι διαφορετικά, πάλι σας λέω, θα, θα, μειωθούν οι πόροι, φοβάμαι, για την πολιτική συνοχή στο όνομα ότι γίνεται έρευνα και ανάπτυξη και τα αποτέλεσματα δεν θα είναι αυτά που θέλουμε όλοι να υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, για τα κινέζικα προϊόντα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, γιατί στην ουσία ερχόταν σε αντίθεση με τα προηγούμενα που είπατε. Πώς ε, δηλαδή θα ε, μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί προς τα κινέζικα προϊόντα, πώς να αλλάξουμε ε, έτσι ώστε να υπάρχει καινοτομία. Να πάω στην επόμενη όμως ομιλητρία, την κυρία Μανέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λανταμπάσο για την παρουσίασή του. Και φυσικά έχει δίκιο ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει καταδείξει την ανάγκη να ενθαρρύνουμε τις ε, επενδύσεις ε, για την ανταγωνιστικότητα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και να υποστηρίξουμε εκείνες που ε, καθυστερούν στην ανάπτυξή τους. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 να εμπλακούν οι τοπικές αρχές. Να πιστήσω όμως την προσοχή σας στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των σχέσεων μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών ε, είναι περιορισμένη αν δεν ξεπεράσουν ε, τα όρια του ρόλου τους ως απλοί εκτελεστές ε, που εφαρμόζουν ξένες ιδέες και αν δεν συνεισφέρουν στο σχεδιασμό των νέων καινοτομιών. Κύριε Φανσαρό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περισσότερο, αλλά απλώς τουλάχιστον να λαμβάνει υπόψη αυτό που ε, κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε κοντά στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, είμαστε πολύ πιο κοντά από ό,τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έλεγα αναφέρατε την ανάγκη για επιχειρηματικά περιβάλλοντα που ευνοούν την καινοτομία. Συμφωνώ πλήρως με αυτό, όμως υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη-μέλη που ακόμα δεν κατανοούν τον σημαντικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις εθνικές οικονομίες και την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα και δεν υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως θα έπρεπε. Πώς λοιπόν σκοπεύετε να πείσετε αυτές τις εθνικές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν εκείνες τις απαραίτητες συνθήκες ε, για να βοηθηθεί αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον και να δοθεί χρηματοδότηση και αρρωγή στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να εξειδικευτούν στην ανάπτυξη, ή στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτό είναι το ένα μου ερώτημα. Το άλλο μου ερώτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής έχει ήδη προχωρήσει προς την κατεύθυνση της προώθησης της καινοτομίας και ήδη έχει δώσει 86 ε, δισεκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα δύο τρίτα ακόμα δεν έχουν κατανεμηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από τον Επιτρόπο και εσάς ποια είναι η εκτίμηση της, ε, των, των αποτελεσμάτων για τη χρήση αυτών των κονδυλίων στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι ίσως ε, συνειδητοποιήσουμε αν είναι χρήσιμο να, να φύγουν αυτά τα κονδύλια από την ε, πολιτική συνοχής ή να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα για να γίνει σωστή η χρήση αυτών των κονδύλιων. Αγαπητοί συνάδελφοι, εφόσον κανείς δεν θέλει να πει κάτι άλλο, να ζητήσω από τον Μικαήλ Λανταμπάσο να σχολιάσει τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια αυτά και τις ε, επικρίσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τουλάχιστον σε κάποια από αυτά. Πρώτον, ίσως ε, φταίω εγώ που δεν είπα ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούμε ή επηρεάζουμε τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Στόχοι 1, 2 και 3 παραμένουν ως έχουν. Αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα άρθρα 4 και 5 του θεματικού ε, καταλόγους ε, του περιφερειακού Ταμείου. Αυτά είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Να γίνουν όλα αυτά μέσω των ταμείων. Το θέμα είναι η τρέχουσα προγραμματική περίοδο η ανακοίνωση να βοηθήσει τις ε, περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες. Δεν επανειδρύουμε, αν θέλετε, τους στόχους, ούτε στρεβλώνουμε τους ε, στόχους. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας σε καμία περίπτωση. Ίσα ίσα που η συνθήκη λέει ακριβώ το αντίθετο. Οι πολιτικές πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι, όπως λέμε, φιλικές προς την συνοχή. Και αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε ένα νέο όραμα για την Ευρώπη, το οποίο το υποστηρίξετε και εσείς την στρατηγική για το 2020. Υπάρχει λόγος για όλα αυτά. Θέλουμε μια αηφορική Ευρώπη για όλους. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει από την αρχή αυτής της διαδικασίας να εξηγήσουμε πώς οι πολιτικές μας, που είναι το ατέρατο του κοινωνικού προπολογισμού, πώς η δική μας πολιτική θα συμβάλλει σε αυτήν την νέα ε, προσπάθεια. Η ανακοίνωση, συνεπώς, εξηγείται σχετικά ή την τρέχουν στο προγραμματικό περίοδο. Δεύτερον, σε καμία περίπτωση, το υπογραμμίζω, δεν προσπαθούμε να πουλήσουμε εντός αγωγικών κάτι σχετικά για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Δεύτερον, σε καμία περίπτωση, το υπογραμμίζω, δεν προσπαθούμε να πουλήσουμε εντό εισαγωγικών κάτι από τι Βρυξέλλε. Να επιβάλλουμε κάτι στι περιφέρειε. Κάτι το οποίο ξαφνικά κάποιοι φάνταστοι υπάλληλοι θέλησαν να φορτώσουν στι περιφέρειες. Το αντίθετο. Η ανακοίνωση προβλέπει μια διαδικασία από τη βάση προς τα πάνω, γιατί οι περιφέρειες γνωρίζουν τι χρειάζονται. Προσπαθούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε με γνώμονα αυτό τους πόρους που διαθέτουν οι Βρυξέλλες για την περιφερειακή ανάπτυξη. Στην οικονομική βιβλιογραφία δεν η οικονομική πολιτική που βασίζεται στην συνοχή δεν λέει ότι χρειαζόμαστε νέε θέσει εργασία από ανταγωνιστικέ επιχειρήσει. Αυτό ακριβώ είναι ο στόχο μα όταν λέμε ότι θέλουμε να προαγάγουμε την καινοτομία. Η καινοτομία βρίσκεται στην καρδιά ακριβώ τη προσπάθεια. Και εδώ προβλέπουμε και την ανακατανομή, αλλά θέλουμε να μεγαλώσουμε ταυτόχρονα και την πίτα έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο να αναδιανύμουμε και ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στον στόχο 1. 80% των πόρων μα πηγαίνουν σε αυτού που του χρειάζονται περισσότερο. Άρα χρειαζόμαστε και καινοτομία, ακόμα και στι απότατε αγροτικέ περιοχέ. Και να πω στον Έλληνα συνάδελφο, προκειμένου ότι είχαμε εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα στο Βόρειο Αιγαίο ε, ή στην Κεντρική Μακεδονία χάρη στα προγράμματα αυτά καινοτομίας. Η καινοτομία αυτα καινοτομια η καινοτομια ειναι κρίσιμη σημασία και θα είναι, είναι υποχρεωτική για τις περιφερειές μας για να δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασία, δραστηριότητες και τελικώ εισόδημα. Και απαντώντα τον κύριο Φανιστελρόη να πω ότι και μάλιστα να ξαναπώ ότι δεν είχα χρόνο ίσω ή δεν, δεν είπα αρκετά καλά η έκθεση ήταν πηγή έμπνευσης και βρίσκεται στο επίκεντρο και αυτή τη δική μου παρουσίαση όσον αφορά την ανάγκη συνεργειών μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων τα οποία είναι διαθέσιμα για την προαγωγή των στόχων της Κομισιόν. Η ανακοίνωση αυτό ακριβώ προσπαθεί να αποδείξει ότι δηλαδή υπάρχουν περιθώρια βελτίωση και ότι υπάρχει ανάγκη για ευρύτερε συνέργειε στο πλαίσιο, στο πρόγραμμα πλαίσιο για την ε, καινοτομία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάλι συγγνώμη δεν το είπα, Μιλάμε για διπλωματευρές τεχνίας, για ψηλή τεχνολογία, μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για μικρές ε, καινοτομίες, για μικρές τροποποιήσεις, βελτιώσεις που δημιουργούν και εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι τα πράγματα που θα μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς, θα δώσουν πλεονεκτήματα και θα κάνουν και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ακόμη πιο ανταγωνιστικές. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο τρίτα των θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε τέτοιου είδου εταιρείε. Και δεν είναι εταιρείε οι οποίε ε, παραδοσιακά συμμετέχουν στο πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία και την έρευνα. Όχι. Ο στόχο μα είναι όμω αυτό. Και αυτά προσπαθούμε να εξηγήσουμε στου πολίτε, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Γιατί υπάρχουν έργα τα οποία είναι απτά, ε, όπω ένα αυτοκινητόδρομο, αλλά υπάρχουν και Άιλες πρόοδοι όπως η κοινοτομία στην έρευνα και που είναι αόρατες για τον Μεσοπολίτη, δεν είναι στα πρωτοσέλιδα ποτέ των εφημερίδων. Το Κοινοβούλιο θέλω να μας βοηθήσει αυτήν την προσπάθεια γιατί δεν είναι εύκολη όπως προείπα. Δεν πρόκειται πάντως για διαστέρευση των αρχικών μας στρατηγικών στόχων. Απλώς χρειαζόμαστε περισσότερη καινοτομία για να τους υποστηρίξουμε. Πιστεύουμε στην καινοτομία Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε καινοτομία Αυτά για τους στόχους. Τώρα συμφωνώ με αυτό που είπατε. Ναι, περισσότερη γνώση, ναι, ανταλλαγή γνώσης. Και έδωσα ίσως περιβολικά πολλά παραδείγματα ακριβώ για να αποδείξω ότι θέλουμε αυτές οι πρακτικές να περάσουν από μια περιφέρεια στην άλλη. Δεν υπάρχει βέλτιστη πρακτική, υπάρχουν καλές πρακτικές, πρέπει να τις κυκλοφορήσουμε και από εκεί πέρα η κάθε περιφέρεια από μόνη της θα προκρίνει τη μέθοδο, την στρατηγική και το ποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα θα χρειάζονται είδου κοινοτομία για να δημιουργήσουν θέσει εργασία. Για να προχωρήσουμε τώρα προς τα εμπρό, από εδώ και πέρα, για περισσότερη συνοχή, χρειάζεται εξή. Καταρχήν, η συνοχή σημαίνει επικέντρωση σε αυτού οι οποίοι αντιμετωπίζουν τι μεγαλύτερε δυσκολίε όσον αφορά την πρόσβαση στο πρόγραμμα πλαίσιο δηλαδή και τις άλλες πολιτικές για αριστεία. Μέσω του μέσου αυτού και του Περιφερειακού Ταμείου οι κυβερνήσεις και οι περιφέρειες, ιδιαίτερα οι πιο φτωχές, θα μπορέσουν να κάνουν βήματα προς τα εμπρός. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ευφύης ανάπτυξη, μιλάμε για γνώση, για γνώση εφορικού χαρακτήρα. Η πολιτική αυτή προάγει την ευφύη ανάπτυξη και έτσι προαγεί την ανάπτυξη της θέσης εργασίας και δει στις ε, φτωχότερες περιοχές που το χρειάζονται περισσότερο. Ποιες είναι τώρα οι συγκεκριμένες προτεραιότητες, ποιος τις ε, ελέγχει, ποιος συντονίζει τα προγράμματα. Στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουμε το περιφέρειες για τη γνώση, περιφέρειες, με συγχωρείτε για την ανάπτυξη κλπ. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις και τις περιφέρειες για να μάθουμε ένας από τον άλλον. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα η οποία θα προάγει την δικτύωση, τις επαφέ, την αλληλοϊποστήριξη. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε τα λεγόμενα fast track δίκτυα. Ήταν στα στήφανες που σας έδειξα, δεν μίλησε πολύ όμως για το θέμα. Είναι χώροι, στρογγυλά τραπέζια αν θέλετε, που γύρω από τα οποία συγκεντρώνονται οι ενδιαφερόμενοι και ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες, προτάσεις. Όμως δεν επιβάλλουμε τίποτα σε κανέναν η συζήτηση γίνεται στο ίδιο επίπεδο, όλοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και μεταξύ τους αποφασίζουν ότι θέλουν. Η κυβέρνηση τώρα, κυβερνήσεις και περιφερειακές αρχές. Είμαστε κοντά στις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές, όντως, ε, και δεν λέμε σε κανέναν ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα. Αντί να τους υποδείξουμε εμείς τους τομείς στους οποίους ε, πρέπει να επενδύσουν, για να του πούμε πώ θα το κάνουν, προσφέρουμε αντιθέτω ένα ευέλικτο στρατηγικό πλαίσιο το οποίο εστιάζει στι διαδικασίες. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω. Προσπάθησα λίγο πριν να εξηγήσω ότι πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκινάει από τη βάση. Από τον ιδιωτικό τομέα και από τους πολίτες. Το ζήτημα είναι πώς θα ξοδέψουμε τα δημόσια κονδύλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πώς θα υλοποιήσουμε την ατζέντα της καινοτομίας. Αυτά μπορούν να γίνουν, αλλά χρειάζονται καλή διακυβέρνηση σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι κυβερνήσει πρέπει να συνεργαστούν και αυτές με τις περιφέρειες και τους δήμους. Αυτό είναι η κατακόρυφη διάσταση. Έχουμε όμω και την οριζόντια διάσταση λέμε όχι στα στεγανά. Ή τα, η, μας πρόταση, αν θέλετε, είναι ότι για να προαχθεί η κοινοτομία πρέπει να συνεργαστείτε, να συνδυάσετε τις προσπαθίες σας. Ούτω ή άλλω και εμεί συνεργαζόμαστε στην Κομισιόν, τέσσερι διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει και τέσσερι επίτροποι. Αξιολόγηση τη αποτελεσματικότητα. Τελευταίο θέμα. Δεν θέλω να αναφερθώ στα ήδη πεπραγμένα, αλλά θέλω να ξέρετε το εξή και το λέει και η ανακοίνωση. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αξιολόγηση και μάλιστα συνεχή διαρκή αξιολόγηση. Και για να γίνει αξιολόγηση απαιτούνται δείκτες. Η πιο πρόσφατη προσέγγιση μας με την κατηγοριοποίηση των εξόδων αρχίζει να βαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Γνωρίζουμε καλύτερα τι κάνουμε, αξιολογούμε καλύτερα, αλλά ακόμη απέχουμε πάρα πολύ από τον στόχο. Δηλαδή, εξαιρετικά εργαλεία αξιολόγησης που μας επιτρέπουν σε διαρκή βάση να βελτιώνουμε τις πολιτικές μας. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε λοιπόν αξιολόγηση. Το λέει αυτό σαφώς η ανακοίνωση και για τις αξιολογήσεις εξαρτώμεθα σε πολύ μεγάλο βαθμό από την βούληση των κρατών μελών να συνεργαστούν με εμά, να καθιερώσουμε βασικούς δείκτε απόδοση για να μετρήσουμε την απόδοση της καινοτομία. Και ναι, δεν είναι μόνο τα διπλώματα είναι οι θέσει εργασία, ε, τα προϊόντα είναι η απασχόληση σε ειδικού τομεί. Προσπάθησα Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, να απαντήσω όσο καλύτερα μπορούσα. Αν έχω ξεχάσει κάτι, παρακαλώ, συγχωρήστε με και να μου το πείτε. Ευχαριστώ, κύριε Νταμπάσο. Όπω βλέπετε, η καινοτομία αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για όλου του συναδέλφου. Ορισμένοι έχουν ανησυχίε στο πλαίσιο τη πολιτική συνοπτικής γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και ιδίως οι φτωχές περιφέρειες ε, ε, θέλουν να δουν την αυξανόμενη σημασία της καινοτομίας γιατί πιστεύουν ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να διατηρήσουν ε, τις βιώσιμες θέσεις εργασίας που δεν θα χαθούν ε, αύριο στα πλαίσια των νέων αναδυόμενων παγκόσμιων οικονομιών. Έτσι λοιπόν, οποιαδήποτε βήματα γίνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη ΓΑΜΑ Region, θα σας θα παρακαλούσαμε να έρχεστε εδώ και να μας κρατάτε ενήμερους για όλα τα βήματα που θέλει να υλοποιήσει η Κομισιόν και επίση να μα ενημερώσετε και τι γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών. Γιατί κατανοούμε ότι κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα ε, αυτή η ανακοίνωση έλαβε πολύ μεγάλη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη. Θα θέλαμε λοιπόν συνεχώ να είμαστε ενήμεροι για τα σχέδιά σα. Σα ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά σα σήμερα στη συνάντησή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 6 τη ημερικής διάταξη. Ε, είναι ένα σημείο ο είναι ο κύριος Φανής Τελρόη. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις για το Ευρωπαϊκό Έτος της 2012. Λαμπέρ, αν θες μπορείς να παρουσιάσεις το σχέδιο κειμένου. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ πρόκειται για ένα θέμα λιγότερο πολύπλοκο από το προηγούμενο. Πρόκειται για ένα θεματικό έτος που θέλει να ενεργοποιήσει και να αφιερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τη μορφή μιας νέας δραστηριότητα. Μιλάμε για μια ομάδα, λένε, και πιο σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην πρώτη θέση παγκοσμίω ό,τι αφορά τη γύρανση του πληθυσμού, αλλά και στις δημογραφικές αλλαγές έχουμε μείωση του πληθυσμού. Αυτό μας οδηγεί στο να προβληματιστούμε. Έχουμε ένα όλο ένα και μικρότερο πληθυσμό και σε αρκετές περιφέρειες ήδη γίνονται ορατά τα αποτελέσματα. Αρκεί να δούμε τη Ρουμανία, την πρώην Ανατολική Γερμανία και ορισμένες ε, γαλλικές περιφέρειες. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση του πληθυσμού. Ήδη Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό σε πολλές ε, συνεδριάσεις ε, και μάλιστα και στη δική μου περιφέρεια. Θέλω να επικεντρωθώ σε τέσσερα σημεία. Καταρχήν πιστεύω ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τον τίτλο αυτού του θεματικού έτους. Θα πρέπει να λέμε ενεργός γύρανση βεβαίως αλλά και να ευνοήσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των ε, γενεών. Δηλαδή δεν μιλάμε εδώ μόνο για τους ηλικιωμένου, αλλά θέλουμε να επιμείνουμε και στην αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των γενεών. Γνωρίζουμε ότι έχουμε όλο ένα και μικρότερο αριθμό ενεργού και στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ σημαντική η ελεγγύη μεταξύ των γενεών. Θα πρέπει να ε, μιλάμε λοιπόν για ενεργογύρανση. Πολύ ωραίο είναι αυτό το θέμα, αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ελεγγύη. Φυσικά όλα αυτά σημαίνουν ότι και οι περιφέρειες πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά με μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μιλώ για ευρωπαϊκά μέσα. Και επίσης ε, έχουμε εδώ και ε, το ρόλο που θα διαδραματίσουν οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών. Δεν έχουμε ακόμη εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρουν αυτές τις τεχνολογίες κάτι ακόμη επί του οποίου δεν επέμενα. Θέλω να θέσω την εξή ερώτηση στους συναδέλφους. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τη χρηματοδότηση. Γιατί να έχουμε ένα ευρωπαϊκό έτος ε, για ένα τόσο φιλόδοξο θέμα χωρίς πόρους για να κάνουμε κάτι απτό, δεν ξέρω αν είναι κάτι θετικό. Σας ρωτώ λοιπόν. Θέτω το ζήτημα των χρημάτων. Δεν θα έπρεπε, το χάρη, να πούμε ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια για ένα τέτοιο έτος και να μην αρκούμαστε απλώ σε ένα μεγάλο επίβολο τίτλο. Δηλαδή να είναι πολύ ενδιαφέροντα θεωρητικά, χάρτη, όλα αυτά που συζητούμε, αλλά να μην έχουμε καμία χρηματοοικονομική δέσμευση. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι θέλουν να ε, να θέσουν και την πτυχή των ε, συντάξεων. Βέβαια, εγώ δεν αναφέρθηκα σε αυτό, ήθελα να περιοριστώ στις γενικέ πτυχέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α δώσουμε τώρα το λόγο στους σκιώδεις ε, εισηγητέ. Κυρία Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει αυτό το σχέδιο για την ανακοίνωση του 2012 για την έτος ενεργούς γύρανσης. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, στο γεγονός ότι θα πρέπει να προσανατολιστούμε προς ε, την τρίτη ηλικία και να ε, αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτής της πληθυσμιακής ομάδας. Ο στόχος είναι να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και τις τοπικές αρχές όπως και την κοινωνία των πολιτών για να υποστηρίξουν και αυτοί με τη σειρά τους την ενεργό γύρανση να κινητοποιήσουμε ε, την ε, ομάδα του πληθυσμού άνω των 55 ετών να δείξουμε αλληλεγγύη. Αυτή η πρόταση λοιπόν επιδεικνύει ε, πώς ακριβώς γίνεται όταν έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Αναφέρει διάφορα θέματα και πτυχές αυτού του ζητήματος. Ως σχεδόν εισηγήτρια λοιπόν χαιρετίζω την ε, μεγάλη εμπλοκή των ε, περιφερειακών αρχών και των τοπικών ε, αρχών. Αν συμφωνήσουμε σε αυτή την θέση, ελπίζω ότι θα την εγκρίνουμε και οι τοπικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να γνωρίσουν καλύτερα το θέμα. Ε, θα ήταν καλύτερα να διευρύνουμε ε, λίγο τον τίτλο, ε, να τον κάνουμε ας πούμε αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Αυτό θα ήταν κάτι πιο σωστό και θα αντιπροσώπευε και το πνεύμα αυτής της πρότασης. Ελπίζω λοιπόν ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα εμπλακούν περισσότερο αλλά θα πρέπει να αναφέρουμε και την τοπική κοινωνία, την κοινωνία των πολιτών, η οποία θα πρέπει και αυτή να παίξει ρόλο, όπως και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ελπίζω να υπάρξουν πολλές ε, παρεμβάσεις που θα δώσουν ιδέες ε, για αυτό το έτος της ενεργούς γύρανσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε θέσει πολύ σημαντικά θέματα και όλοι νομίζω συμφωνούμε για τη σημασία που έχει αυτό το ζήτημα. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Να πω ότι στην πέμπτη έκθεση συνοχής ε, που ε, δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες αναφέρθηκε η γύρινση και οι προκλήσεις ε, που προβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλό πως σε αυτό το επίπεδο έχουμε συνειδητοποιήσει τις προκλήσεις που υπάρχουν και ότι μέσα από την πολιτική συνοχή ε, προσπαθούμε να ανοίξουμε αυτή την κλειδαριά. Ε, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το ρόλο των ε, πόλεων στην εφαρμογή και είναι καλό να αναφέρουμε τους εθνικούς συντονιστές οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο του ελεγκτή και του επόπτη ε, της εφαρμογής αυτής της πολιτικής συνοχής. Τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανταλλαγή καλών πρακτικών για παράδειγμα, κάποιες περιφέρειες ε, έχουν ήδη αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα γύρανσης, έχουν ήδη εφαρμόσει καλή διακυβέρνηση, καλές ε, πρακτικές. Επίσης αναφέρθηκε η οικονομική υποστήριξη. Νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί και αυτό το θέμα. Ε, ίσως ε, να υπάρχει δυνατότητα ε, για περαιτέρω χρηματοδοτική υποστήριξη αυτού του έτους, αλλά γενικά να δούμε τι γίνεται με την πολιτική συνοχής. Πώς η συνοχή θα συμβάλλει σε αυτό το τομέα. Επιπλέον, η γύρανση θέτει προκλήσεις και στις υπηρεσίες υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε αν τα κοινωνικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα μπορούσαν να απελευθερώσουν πόρους για αυτόν τον τομέα. Γενικά βέβαια είμαι ικανοποιημένη με την έκθεση και θεωρώ ότι η συγγήτρια, ο εισηγητής μάλλον έχει παρουσιάσει με πολύ σωστό τρόπο όλα τα θέματα που άπτονται αυτού του ζητήματος. Ευχαριστώ δύο οι ομιλητές που ακολουθούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον ε, νέο συνάδελφο, Φανίλη Στελρόη, για την ε, δουλειά του, για την ενεργογύρανση. Νομίζω ότι το θέμα της ενεργογύρενσης είναι πάρα πολύ σημαντικό εγώ στη Γαλλία έχω εκλεγεί σε ένα γενικό συμβούλιο που είναι το αρμόδιο επίπεδο για την αρρωγή στους ηλικιωμένους και στα άτομα με δυσκολίες. Και ήδη έχουμε το 60-65% του τίσου υπερπολογισμού μας να αφιερώνεται εκεί. Δηλαδή, όταν μιλάμε για χρηματοδοτικά μέσα, νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλο και περισσότερου πόρου για να διαχειριστούμε όλη αυτή την προβληματική. Το Ευρωπαϊκό Έτο τη Ενεργού Γύρανση έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις προσπάθειε των κρατών μελών και τη τοπική αυτοδιοίκηση, των κοινωνικών εταίρων αλλά και τη κοινωνία των πολιτών για να αξιοποιήσουν καλύτερα το δυναμικό των ε, ηλικιωμένων ατόμων που είναι ακόμη στην αγορά εργασία. Έτσι λοιπόν ε, πιστεύω ότι με την πρωτοβουλία αυτή τη Κομισιόν θα επιτρέψουμε στου ηλικιωμένου ε, να καταπολεμήσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να αξιοποιήσουν καλύτερα το έργο Του Ξέρουμε ότι όλοι πρέπει να εργαζόμαστε, το λένε και περισσότερο, γι' αυτό άλλωστε στη Γαλλία κάνουμε και την μεταρρύθμιση του εξωτερικού συστήματο. Εμείς ε, τα καταφέραμε τελικά, αν και ήταν δύσκολο και πιστεύω ότι είναι σημαντικό και οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν ένα δικτύο βέλτιστων πρακτικών για την ενεργοκίνηση. Η ένταξη των ε, ηλικιωμένων εργαζομένων είναι σημαντική πτυχή για την κοινωνική αλλά και την εδαφική συνοχή. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ. Thank you, ε, Ευχαριστώ κυρία Αντιπρού. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν ε, θα ήθελα να συμφωνήσω όπως είπε ο κύριος ε, Φανής Τελρόη με το να συνεισφέρουν οι πιο ηλικιωμένοι στην κοινωνία δυστυχώς πολύ συχνά σε αυτή τη συζήτηση για τις δημοκρατικές προκλήσεις ε, φαίνεται να παρουσιάζει τους πιο ηλικιωμένους ως άχθος και όχι ως ενεργό πόρο για την κοινωνία και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό εδώ. Εγώ καλωσορίζω λοιπόν απόλυτα την πρόταση του να προσθέσουμε και την προώθηση της ε, διαγενολογικής αλληλεγγύης στον τίτλο Ξέρω ότι στην Ισπανία, από την Ισπανική Προεδρία, έλαβε χώρα μία διάσκεψη όπου τονίστηκαν πολλές σημαντικές πτυχές ε, σχετικά με την ενεργογύρανση και τι σημαίνει η αλληλεγγύη μεταξύ των ε, γενεών και η κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, και η σχετική πλατφόρμα για την κυβέρνηση παρουσίασαν εκεί διάφορες ιδέε σε σχέση με το τι θα ήταν απαραίτητο σε ό,τι αφορά τώρα την πρόθεση της διανολογική αλληλεγγύη. Υπάρχουν κάποια πολύ καλά σχέδια στη δική μου εκλογική περιφέρεια που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο με τη χρήση σχετικά λιγοπόρων και ξεπερνάμε το θέμα της αλληλεγγύης που πρέπει να επιδεικνύουμε εν ώψη των δημογραφικών ελλαγών. Εκεί έχουμε και το πώς θα φέρουμε κοντά τους νέους με τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους μέσα σε οικογενειακές δομές που έχουν αλλάξει σήμερα ε, γιατί σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο φυσικός τρόπος της της ε, αλληλεγγύης μεταξύ των γενναιών που υπήρχε παλιά. Ε, πολλές ε, φορές βλέπουμε ε, μάλλον αυτά τα, τα project έχουν να κάνουν πολλά με τους νέους που δεν κάνουν τίποτα και στεκόνται στο δρόμο ή παίρνουν ή κάποια άλλα ασχολούνται με τους ηλικιωμένους. Ε, επίσης ε, έχουμε και συναντήσεις όπου συμμετέχει και ο εκπρόσωπος των ηλικιωμένων. όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί το είπε και ο κ. Φενιστερόη. Αυτά τα θεματικά έτη ε, μπορούν να ακολουθήσουν μια-δυο οδούς. Ε, καταρχήν, ε, το θέμα είναι να μην έχουμε απλώς κάτι επί χάρτου και παρά μόνο μια-δύο συναντήσεις. Να έχουμε και κάτι πρακτικό, αλλά μπορεί να έχουμε και μια δεύτερη οδό, δηλαδή να αποτελεί αυτό μια βάση για την υλοποίηση εργασίας. Παίρνουμε το χάρη, το έτος που είχαμε για τα άτομα με αναπηρία, συλλέχθηκαν ένα εκατομμύριο υπογραφές και έτσι προωθήθηκε μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια για την οδηγία για την ισότητα πέραν, πέραν της ε, απασχόλησης. Έτσι λοιπόν αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για νέους τρόπους εργασίας και νομίζω ότι η ευκαιρία να έχουμε το 2012 αυτό το θεματικό έτος κατόπιν ε, του φετινού θεματικού έτους ε, που είναι για την ε, καταπολέμηση της φτώχειας και έχουμε και το 2013 το έτος του ελληνισμού θεωρούμε ότι μπορεί να είναι αυτό το έτος όπου με διάφορα συγκεκριμένα προγράμματα μπορούμε να δώσουμε ουσιαστικά πρόθεση σε διάφορα σχέδια που θα υιοθετηθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Ήθελα να πω ότι εδώ ο τίτλος αναφέρεται στην ενεργό γύρανση. Καλώς είναι. Και εδώ τείνουμε να βλέπουμε ε, το θέμα αυτό πέραν της συνταξιοδότησης γιατί αν δούμε τον τίτλο έχει, ισχύει για όλους και μάλιστα ο όρος active ενεργός αντίκειται στον όρο inactive ενεργός και αυτό έχει να κάνει με όλες τις γενιές και κυρίως δεν μιλάμε για τη σωματική δραστηριότητα, τη φυσική δραστηριότητα, γιατί προσπαθούμε να αναπτύξουμε για κάποια μέτρα και για την φυσική δραστηριότητα και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να είναι ενεργοί σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Αυτό θα εφελίσει τον τρόπο που ζουν γενικότερα. Αυτό είναι πλεονέκτημα για την κοινωνία, ενώ η αδράνεια οδηγεί σε πάρα πολλά προβλήματα και σε προβλήματα υγείας. Έτσι λοιπόν καταρχήν και πρέπει να επικεντρωνόμαστε. Δεύτερον, το όλο ζήτημα του να έχουμε ε, ενεργό γύρανση, δηλαδή να έχουν δραστήρια γυρατιά οι άνθρωποι, αυτό σημαίνει ότι όταν ε, εγκαταλείπουν την εργασία τους ε, θα μπορούν το χάρη να ταξιδεύουν ή να κάνουν άλλες δραστηριότητες και επίσης υπάρχει και πανητεραστή δυνατότητα να επικεντρωθούν στον εθελοντισμό. Και αυτό είναι μια επιλογή τρόπου ζωής μάλλον. Δεν ξεκινάω όταν συνταξιδοτηθεί, αλλά θέλω να εστιάσουμε περισσότερο λοιπόν σε δραστηριότητε που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωή και τι σχετικέ επιλογέ που οδηγούν σε μια πιο υγιεινή ζωή, παρά σαν κάτι που θα ξεκινά από τα 65 και άνω. Και εδώ συμφωνώ με το Λάμπερτ, αν έχουμε το έτος της κοινωνικής ένταξη, το έτος της ενεργού γύρανσης και το έτος του εθελοντισμού σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα για όλα αυτά τα έτη και πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πιλωτικά προγράμματα που θα αναπτυχθούν. Γιατί θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς στο τέλος κάθε έτους ε, πόσοι πολίτες γνώριζαν ότι είχαμε συγκεκριμένο ε, θεματικό έτος και τι αντίκτυπο είχε. Και νομίζω ότι έτσι θα συνεχιστούν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Πριν να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Φανστερό για τα τελικά σχόλια, κύριο Φανμάτσεκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος μάλλον Μάτσεκ, ε, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στην ερώτηση για τον προπολογισμό. Η Κομισιόν δεν έχει προτείνει συγκεκριμένο προπολογισμό για αυτό το θεματικό έτος, το συγκεκριμένο, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε πολλέ δραστηριότητε από υφιστάμενε γραμμέ προπολογισμού και ευκαιρίε χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν θα έχουμε κάποιους πόρους ε, για την εκστρατεία ενημέρωσης ε, και αυτό είναι το κύριο εργαλείο για το ευρωπαϊκό έτος και κατόπιν έχουμε πολλά προγράμματα. Ήδη σήμερα μέσω αυτών μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε σχετικές δραστηριότητες με την ενεργό και έχουμε συναντήσει τρεις φορές και με συναδέλφους από άλλες γαμαδέλτα και προσπαθούμε να ε, ε, θέσουν και αυτοί ως προτεραιότητα την ενεργό γύρανση στα υφιστάμενα προγράμματα. Δηλαδή αυτό ισχύει ήδη. Έχουμε πολλά προγράμματα όπως διαβίωμα άθηση κτλ. Που, όπου ήδη γίνεται αυτό, αλλά θέλουμε το 2012 να οργανώσουμε και τήσιες ε, συναντήσεις που θα λαμβάνουν χώρα για την ενεργό και από τη ΓΔ απασχόληση αλλά και σε άλλες ΓΔ. Μη φοβάστε λοιπόν, θα υπάρχουν δραστηριότητε και υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, αλλά διαφέρει η κατάσταση από το 2009 που είχαμε το έτος ε, για την δημιουργικότητα και την καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φανίστερο, θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, για τις παρεμβάσεις σας. Νομίζω ότι οδεύουν προς την κατεύθυνση τα σχόλιά σας και μου επιτρέπουν να εμπλουτίσω το κείμενο. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στήριξη για την εκθεσή μου. Πιστεύω ότι θα επιμείνουμε στα γεγονότα, γιατί Κατά το πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτους η Κομισιόν ε, θα μας παρουσιάσει συγκεκριμένες ε, προτάσεις για το ζήτημα αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε ε, κάποιο χρόνο στη θέση μας στις 18 Δεκεμβρίου, ίσως λίγο περισσότερο χρόνο χρειαστεί για τις τροπολογίες. Τώρα, για τη χρηματοδότηση, για τα κονδύλια. Συμφωνώ με την Κομισιόν να χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους πόρους, αρκεί να είναι για απτά προγράμματα, να είναι, μιλάμε για κάτι ξεκάθαρο. Δηλαδή να μην ε, ξαναπέσουμε στη γραφειοκρατία. Αλλά σε αυτά τα διάφορα προγράμματα που αναφέρετε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Διαφορετικά δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε επί της προσέγγισης που θα ακολουθήσουμε. Αν στην αρχή του επόμενου έτους διαπιστώσουμε ότι όλες οι προτάσεις οδεύουν προς την κατεύθυνση, δεν θα προτείνω άλλες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το μόνο που πρέπει να αποφασίσουμε τώρα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Είναι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίας ανοιχτή κατάθεση για να γίνει η ψηφοφορία το Γενάρη. 8 Δεκεμβρίου, λοιπόν, 6 μετά μεσημβρία είναι η προθεσμία. Να πάμε τώρα στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Οι Ιρλανδοί συνάδελφοι πριν από λίγο καιρό μας ζήτησαν να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μας ενημερώσει και να γίνει μια σύντομη αναλλαγή απόψεων για το πρόγραμμα PIS. Έχουμε σήμερα την κυρία Ανιές Λίντερμανς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. παρόλο που υπάρχει όλο αυτό ο θόρυβο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια φυσιολογική συζήτηση. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Λίντερμαν για να μας δώσει κάποια στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα PIS. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι μου δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσω την Επιτροπή σας για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαδικασία ε, ειρήνευσης ε, το πρόγραμμα PIS στην Ιρλανδία. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης PIS είναι η πιο ξεκάθαρη εκδήλωση της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία. Έχουμε συνεισφέρει 1,3 δις ευρώ μέσα ε, σε τρία προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν το 1994 και Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 349 εκατομμύρια από το 1989. Θα επανέλθω αργότερα στην οικονομική ε, συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω όμως ότι η ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία υποστηρίχθηκε και μέσω άλλων μέσων μη οικονομικών. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Βαρόσο, ήταν ο πρώτος ε, ξένος αξιωματούχος, ο οποίος πήγε το Μάιο του 2007 για πρώτη φορά στην περιοχή, μετά από τη συμφωνία ε, που έγινε εκεί. Μετά ε, δημιουργήθηκε μία task force στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα βοηθήσει την Βόρεια Ιρλανδία να χρησιμοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να περάσει για να έχει μια ομαλή μετάβαση στην ειρήνη. Να σας ενημερώσω ότι στο αποτέλεσμα των εργασιών της Task Force η Βόρεια Ιρλανδία μπόρεσε να εμπλακεί περισσότερο στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Υπάρχει ανταλλαγή εξωματούχων, ε, και ξεκινάμε από αυτό ε, και φτάνουμε μέχρι ε, μια μεγαλύτερη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πολιτικές, στα διευρωπαϊκά δίκτυα και το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Όπως ανέφερα, η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία εκφράστηκε και με οικονομικούς όρους μέσω δωρεών στο Διεθνές ε, Ταμείο για την Ιρλανδία από το 1989 και μετά και μέσω από το πρόγραμμα Peace ε, που είναι ε, ένα πρόγραμμα των διαρθρωτικών ταμείων. Τον Απρίλιο φέτος ήμασταν για πάλι εδώ στην Επιτροπή σας για την έκθεση του κυρίου Σονκέλη για τον κανονισμό Κοινοβουλίου Συμβουλίου σχετικά με τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την ε, Ιρλανδία ε, περίοδος 2007-2010. Η έκθεση τότε, μεταξύ άλλων, έδινε ε, πολύ θετικούς τόνους ε, για το αποτελέσμα της εργασίας αυτού του ταμείου και ανέφερε την ανάγκη να συνεχιστούν τέτοιες πρωτοβουλίες. Επίσης υπήρχε η έκθεση δύο πρωτοβουλίας τη κυρίας Ντεμπρά σχετικά με την ευρωπαϊκή υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Βόρειο Ιρλανδία, όπου ανέφεραν και πάλι οι συνάδελφοι θετικά σχόλια για το θέμα αυτό. Επίσης, έκθεση πρωτοβουλία τη Επιτροπής ε, Κοινωνικών Υποθέσεων να έχει τα ίδια θετικά σχόλια. Επίσης, ανεξάρτητες ε, αξιολογήσεις από την διοικητική αρχή του ε, προγράμματος ΠΙΣΕ και του Ταμείου αναφέρουν ποιος είναι ο θετικός αντίκτυπος αυτών των παρεμβάσεων. Σε όλες αυτές τις αξιολογήσεις αναφέρεται ότι ε, η ειρήνη και η συμφιλίωση είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία η οποία θα πρέπει ε, συνεχώς να υποστηρίζεται με τέτοιες παρεμβάσεις. Θα πρέπει νομίζω να σας αναφέρω κάποια νούμερα. Από την αρχή του το Ταμείο για την Ιρλανδία ε, έχει δώσει πάνω από 830 εκατομμύρια σε πάνω από 600 προγράμματα σε όλο το φάσμα υποστήριξης 1,4 δις για κάθε λίρα που επενδύθηκε και 2,2 επιπλέον από, άλλες, από άλλους πόρους. Συνολικά δηλαδή υποστηρίξαμε 55.000 θέσεις εργασίας. Επίσης υπάρχει συνδυασμένος προϋπολογισμός πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ και πάνω από το 1,1 ε, εκατομμύριο, δισεκατομμύριο είναι συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χρηματοδοτήθηκαν 12.000 προγράμματα και δημιουργήθηκαν 2.000 θέσεις εργασίας όπως ε, εκπαιδεύτηκαν και πάνω από 9.000 άτομα. Το PIS 3 έδωσε 333 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 225 προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Όσο εντυπωσιακά και να είναι αυτά τα νούμερα, ο αντίκτυπος ε, του ΠΙΣ και του Ταμείου πάει πέρα από τους ποσοτικούς δείκτες. Είναι οι ποιοτικοί δείκτες που δείχνουν καλύτερα την εικόνα σχετικά με την ειρήνη και τη συμφιλίωση να μερικά παραδείγματα. Οι παρεμβάσεις ε, του Ταμείου στην Βόρεια Ιρλανδία συνεισέφεραν στην ε, ολένα και μεγαλύτερη ενεργό δράση των, των δύο κοινοτήτων και στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ αυτών. Ε, όλα αυτά τα εργαλεία βοήθησαν να διατηρηθεί ο ρυθμός ε, προόδου όταν ήταν αργή η πολιτική ε, πρόοδος. Ε, ακόμα και όταν οι δύο κοινότητες ε, δεν μιλούσαν μεταξύ τους, η χρήση αυτών των μέσων ήταν ο μόνος τρόπος να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να πάρουν από κοινό αποφάσεις. Και τα δύο ταμεία στην ουσία πήγαν στις ρίζες του προβλήματος και βοήθησαν τον κόσμο να, να βρει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τα θετικά της ε, ειρηνευτικής διαδικασίας. Επίσης ε, έγινε αποδεκτή η διασυνοριακή συνεργασία μέσω αυτών και έγινε, το... έγινε φυσιολογική. Επίσης, ε, οι τρεις, τα τρία ενδιαφερόμενα μέρη εμπόρεσαν να συμμετέχουν από κοινού και αυτό ε, έδωσε την εντύπωση στον κόσμο ότι είχαν και αυτοί να προσφέρουν κάτι. Γενικά υπήρξε μία ε, εμπειρία σχετικά με τον τρόπο που, που εκτελείται μία ειρηνευτική διαδικασία. Οι εκθέσεις, ε, οι δύο πρωτοβουλίες και οι άλλες εκθέσεις έχουν αναγνωρίσει αυτές τις εμπειρίες. Το πρόγραμμα PEACE ε, έχει δημιουργήσει ένα, ένα δίκτυο ειρήνευσης μέσα από το οποίο ε, δίκτυα και οργανώσεις από την Ευρώπη και πέραν αυτής μπορούν να συμμετάσχουν. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη δημιουργία της ειρήνης αλλά και των τοπικών αρχών για τις πρωτοβουλίες ε, συμφιλίωσης είναι δύο από τα εργαστήρια που βοήθησαν μέσα από αυτό το δίκτυο. Να τελειώσω αναφέροντας κάποια λόγια σχετικά με το μέλλον του ΠΙΣ και του IFI, του Ταμείου για την Πορειρλανδία. Το IFI έχει αποφασίσει το 2006 να μην ζητήσει νέα χρηματοδοτική συνεισφορά από ε, δωρητές ε, στην περίοδο μετά από φέτος. Ε, Παρ' όλα αυτά, επειδή αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά, ε, δεν θέλει να σταματήσει τις δραστηριότητες του και τα κράτη-μέλη της ε, Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησαν από την Κομισιόν να σκεφτεί αν θα μπορέσει να συνεχίσει την χρηματοδότηση μια σειράς περιορισμένων στοχευμένων δραστηριοτήτων. Ε, η Κομισιόν εκτιμά τη δουλειά των, του Ταμείου και του προγράμματος και ζητά από εσάς ε, να δούμε πώς θα δώσουμε χρηματοδοτική υποστήριξη σε αυτά για την περίοδο 2010-2013 μέσα από τις χρηματοοικονομικές ε, προοπτικές. Επίσης, ε, για την περίοδο μετά το 2013 θέλουμε να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια της συζήτησης των νέων προγραμματικών περιόδων για, το για τα πολιετή προγράμματα. Ευχαριστώ λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας για τη συζήτηση και τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. μπορούμε. Ευχαριστώ την ε, κυρία Λίντεμαν για την ενδιαφέρουσα εισήγηση και για τα καλά λόγια που είπε όχι μόνο για το πρόγραμμα αλλά και για την έκθεση μου πρωτοβουλία στην οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Με την ευκαιρία ένα μεγάλο ευχαριστώ και προς την πρόεδρο μας την κυρία Χούμπνερ η οποία ως επίτροπος διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο αποφασιστικό ρόλο ήρθε η ίδια επιτόπου και είδε πως υλοποιείται το πρόγραμμα και τι ωφελήματα είχε η κυρία Χούμπνερ όμως επιπλέον δρομολόγησε και συνεργάστηκε με την λεγόμενη Barroso Task Force, έτσι όπως τη λέγαμε στην περιοχή μου, στην εκλογική μου περιφέρεια. Και έτσι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα υλοποιήθηκε με επιτυχία. Αξίζει το κόπο νομίζω στο σημείο αυτό να ρίξουμε λίγο ματιά στο πρόγραμμα. Διότι μέχρι το 9 τις τελευταίες ευρωεκλογές το θέμα όταν τρέχουν και παρερχόταν στις σχετικές συζητήσεις και στην Επιτροπή αυτή. Θυμίζω όμω ότι η Επιτροπή μας συμφώνησε να επισκεφθεί τις ε, επαρχίες της ε, Μεθορίου αλλά και άλλες για να δει ακριβώς πώς αξιοποιήθηκαν τα κονδύλια τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής και των περιφερειακών ταμείων. Τώρα, επειδή κάποιοι βουλευτέ δεν είναι εδώ, κάποιοι καινούργοι ήρθαν, καλό θα ήταν να κάνουμε μια ανασκόπηση. Το πρόγραμμα βοήθησε τα θύματα της σύγκρουσης να εμπλακούν στην διαδικασία ειρήνευσης και να προχωρήσουν προς τα μπρος. Δημιουργήθηκε ένα καλό κλίμα το οποίο επέτρεπε πράγματα που ήταν στο παρελθόν αδύνατα και όπως είπε και η κυρία Λίντεμανς ήταν και πάλι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίστηκε ξεκίνησε από τη βάση περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά, τους επέτρεψε να συνεργαστούν στο πλαίσιο κοινών προσπαθειών, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Και εν τέλει απέδειξε ότι τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν να έχουν αποτελέσματα, να παρέχουν υπηρεσίες, να λύνουν προβλήματα. Και αυτό έγινε και με τις δύο πλευρές της Μεθορίου, με δύο διαφορετικές κοινότητες, κάτι το οποίο στο παρελθόν και πάλι ήταν προβληματικό λόγω των γνωστών γεγονότων. Θέλω να τονίσω ότι με όλη μου την καρδιά συμφωνώ με αυτό το οποίο ακούστηκε ότι η συμφιλίωση είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί πολύ χρόνο. Γι' αυτό εμεί είμαστε υπέρ του προγράμματος και θέλουμε να δώσουμε κάτι, να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια, να υπάρχουν ωφελήματα για όλους. Οι οργανώσεις και οι φορείς απέδειξαν την αξία τους ε, στην Ιρλανδία, στα Δυτικά Βαλκάνια και σε άλλες περιοχές του κόσμου μετά από συγκρούσεις. Λοιπόν, μαθαίνουμε και στην περίπτωση αυτή πιστεύω ότι για την σταθερότητα γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα σύνορά μας αλλά και εκτός στα κράτη-μέλη που θα γίνουν κάποια στιγμή στα κράτη που θα γίνουν κάποια στιγμή μέλη θα Αξίζει να μάθουμε πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός ε, για την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Κυρία Λενιμάνς, τα είπε πολύ καλά. Ήσασταν ίσως ε, λίγο πιο αισιόδοξοι το IFI σε σχέση με το PIS 4. Γι' αυτό θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια. Σον. Μπάρμπρα, νομίζω τα είπε, συμφωνώ. Ήδη είναι από την και έχει από πρώτο χέρι εμπειρία και από το κακό παρελθόν και ευτυχώς και από τις καλές ημέρες που ελπίζω θα συνεχίσουν. Δεύτερον, είναι κρίμα που δεν το συζητάμε όλο αυτό στο Κοινοβούλιο γιατί θα το με ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει αν θέλετε την καλή της πλευρά και να την προβάλλει. Οι ορισμένοι έχουν την εντύπωση ότι είμαστε η χειροτερή μηχανή, ο χειροτερός μηχανισμός δημοσίων σχέσεων στον κόσμο. Ακόμα και να κάνουμε κάτι καλό, δεν το προβάλλουμε και αφήνουμε το πεδίο ελεύθερο για τους επικριτές μας. Αν ρωτήσετε τους περισσότερους στην Ιρλανδία ή στον Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος χρηματοδοτεί την ειρηνευτική διαδικασία και τα πρόγραμματα των τελευταίων χρόνων, οι περισσότεροι θα σας πούν <laughs> οι δύο κυβερνήσεις και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Κανείς δεν ξέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει λεφτά. Μάλιστα είναι βέβαιο ότι, ακόμα πιο βέβαιο, ότι δεν ξέρουν ότι είμαστε μεγαλύτεροι δωρητέ. Δεν είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να διαφημίσουμε το πρόγραμμα. Ως ε, εισηγητής θα ήθελα να πω ότι πρέπει να αποδώσουμε φοροτιμής στον Τσιριδέ στον Μάρτιν Μακένες, στην Μπάρμπαρα, σε... στον Ιαν Πέισλι, το πρώην μέλο του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θα ήταν αδιανόητο χωρί αυτούς οι άνθρωποι στην Ιρλανδία, στην Ιρλανδία, να καθίσουν γύρω από το τραπέζι και να δουλέψουν υπέρ της ειρήνης. Φυσικά αυτό δεν ισχύει για μια επικίνδυνη μειονότητα, η οποία υπάρχει ακόμη και σήμερα. Πάντω η ε, ηγεσίε του Σινφέιν, ο Εν Πέισλι, οι συνεργάτε του, είναι άνθρωποι στου οποίου οφείλουμε πολλά. Ο Εν Πέισλι πέρασε χρόνια εδώ. Τον στρογγύλεψαν, τον μαλάκωσαν. Και το λέω αυτό διότι θεωρείται πόσο ο νούμερο ένα Εχθρό. Άλλαξε όμω και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτό. Πήγα στην ε, Βόρεια Ιρλανδία στις 6 Νοεμβρίου πριν από λίγε εβδομάδες. Και πήγα και είδα την υλοποίηση έργων στον Belfast, παράδειγμα, πήγα σε περιοχέ όπου δεν θα μπορούσα κάνει να, να πατήσω σε, πριν από χρόνια γιατί θα ήταν απλώς πολύ επικίνδυνο. Πήγαμε στο Orange Hall όπου μας α, ε, καλωσόρισαν μέλη της άλλης πλευράς όπως α, ε, λέγαμε τον, της Union και συνήθισα με δασκάλους από τα καθολικά σχολεία, από τα Προστατικά σχόλια και αυτή η συνύπαρξη ακριβώ είναι απόδειξη τη πρόοδου που έχει επιτευχθεί. Αξίζουν συγχαρητήρια σε πολλού. Πάντω, υπάρχουν επεισόδια, υπάρχουν ε, διαφωνίε. Ε, Ένα λόγο παραπάνω λοιπόν να συνεχιστεί το σχέδιο αυτό. Όσο περισσότερο διαρκεί η ειρήνη, τόσο λιγότερο πιθανό γίνεται να επιστρέψουμε στις παλιές κακές ημέρες. Ιδιαίτερα σε καιρούς οικονομικής κρίσης υπάρχουν τόσοι νέοι άνεργοι τους οποίους θα στοχεύσουν αυτοί οι οποίοι δουλεύουν υπέρ της βίας. Ένας άλλος λόγος, επαναλαμβάνω, να διατηρηθεί το πρόγραμμα, να συνεχιστεί το πρόγραμμα για την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πρέπει επίση τέλος να διαφημίσει τον ρόλο της ο οποίο ε, την χάνει ακόμη παντελώ άγνωστο για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ευχαριστώ. James Nicholson. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ εσάς και ως Επίτροπο υπογραμμίζω για το πει 3. Σημείωσα ότι η κυρία Λίντεμαν αναφέρθηκε στο σχόλιο του κυρίου Μπαρόζο στην Ιρλανδία. Είναι καιρό κάποιο ανώτατο αξιωματούχο να έρθει στην Ιρλανδία και να συναντήσει και του ε, τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την περιοχή. Ποτέ δεν διαβουλεύτηκε κανεί με εμά. Ε, μόνο ίσω περιστασιακά και στο περιθώριο. Δεν ε, θέλω να με μισημερώ αυτή τη στιγμή, αλλά Όλοι ακούνε για τον Τζέρι Adams και τον Ιαν Πέισλι. Δεν είναι οι μόνοι που δούλεψαν για την υπόθεση. Ο Ζακ Τελόρ ήταν ένας από αυτούς. Ο Τζον Χιούμ, ο Πέισλι και εγώ πήγαμε στο γραφείο του Τελόρ το 1994 και ξεκινήσαμε το πρόγραμμα Peace. Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε ακριβώ να πάνε λεφτά στη βάση, στους ανθρώπους, όχι σε οργανώσει στην κορυφή. Αυτό τότε ξεκίνησε με τον Τελόρ. Δεν πιστεύω ότι η Task Force κατάφερε αυτό που έπρεπε. Υπάρχει ακόμη ένα χάσμα και έλλειμμα υλοποίησης. Και η καθυστέρηση δεν είναι μηνών, είναι ετών. Και αν θέλετε να μάθετε, πηγαίνετε να ρωτήσετε πόσο γρήγορα υλοποιείτε το πρόγραμμα. Μιλήστε με τι τοπικέ οργανώσει, μιλήστε για τη γραφειοκρατία, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην περιοχή. Μιλήστε λοιπόν με αυτού που ξέρουν πραγματικά την κατάσταση. Επίση, οι ομάδε γυναικών στην Βόρειο Ιρλανδία. Και αυτέ αγνοήθηκαν. Μου λένε ότι κανεί δεν ζήτησε τη γνώμη του στο πλαίσιο τη διαδικασία και του πρόγραμματο ποιης. Ύστερα υπήρχε πρόταση 20 εκατομμύρια θα πάνε σε ένα έργο για τις φυλακές 8% του έργου. Εγώ διαφωνώ 100%. Καμία σχέση με, την, με το χρήματα για τους ανθρώπους, για τις οργανώσεις βάσης. Καμία σχέση. Δεν ξέρω λοιπόν αν το πρόγραμμα αποδίδει, αν τα λεφτά πηγαίνουν σε αυτούς που πρέπει. Και ύστερα το πρόβλημα δεν ήταν ότι δεν μιλούσαμε. Εγώ είμαι από ένα χωριό. Οι γείτονέ μου είναι όλων των δογμάτων, όλων των θρησκειών. Μιλάμε μαζί, ξεροζόμαστε, βγαίνουμε. Ακόμα και στι πιο δύσκολε εποχέ. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα και κάτι πρέπει να γίνει. Όμω σε άλλου τομεί πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη. Και δεν ξέρω αν η Μπάρμπαρα θέλει να το κουβεντιάσουμε κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω αν αυτό ε, είναι πρόβλημα των Βρυξελών, τη Ιρλανδία ή του SEUPP που είναι το επιτόπου όργανο, αλλά σίγουρα υπάρχει πρόβλημα υλοποίηση. Μπάρμπερα, και όταν λέγαμε πριν από λίγε μέρε είναι τρομερό ότι οι Υπουργοί Οικονομικών, έχω την εντύπωση, δεν έχουν ιδέα για το πρόγραμμα που πηγαίνουν τα χρήματα και ποιες είναι οι δυνατότητες. Πρέπει λοιπόν να το ξαναδούμε. Το να επενούμε ένα τον άλλον και να λέμε ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά δεν είναι ωφελή. Οι άνθρωποι στην Ιρλανδία πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο. Είπε ο συνάδελφος ότι δεν έχουμε επενδύσει υπερκώς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφωνώ στην Βόρεια Ιρλανδία ξέρουν ότι κάνει πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ξέρουν. Ξέρουν ότι βοήθησε σε δύσκολε εποχέ. Και ξέρουν επίση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμπλέκεται και στι τοπικέ υποθέσει. Λοιπόν, ο κόσμο ξέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, ήρθε η ώρα να ξαναδούμε το πράγμα, να δούμε πώ λειτουργεί το πρόγραμμα, πού υπάρχουν καθυστερήσει, γιατί υπάρχουν προβλήματα, γιατί μια τεράστια γραφειοκρατία εμποδίζει την υλοποίηση γιατί σε μερικές περιπτώσεις έχουμε καθυστερήσει 12-13 μήνες έως και 2 χρόνια. Αυτό είναι απαράδεκτα αργό. Η θέση μου λοιπόν θα ήταν να θέσουμε λοιπόν το ερώτημα στα σοβαρά. Ας μην το λέμε ειρηνή το πρόγραμμα εάν δεν διασφαλίσουμε ότι πράγματι πετυχαίνουμε το στόχο μας. Για ρωτήστε τις ε, τοπικέ αρχέ στην Ιρλανδία, που πήγαν τα χρήματα και ποιο νομίζουν ότι είναι ο στόχο, Εγώ πιστεύω ότι και οι άνθρωποι επιτόπου δεν ξέρουν τι μπορούν να κάνουν με τα χρήματα αυτά. Ύστερα οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απ' έξω. Κανείς δεν τους συμβουλεύτηκε. Κανείς δεν του μίλησε. Θα λέγα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μέσω τη Επιτροπή μα, Ακόμα και αν δεν με πιστεύετε, πηγαίνετε να δείτε επιτόπου τι γίνεται. Εγώ θέλω να τα πω αυτά. Ή δεν μασάω τα λόγια μου. Μιλήστε με τι ομάδε, μιλήστε με τι οργανώσει, οι οποίε δεν ξέρω αν τελικά βλέπουν έστω και ένα ευρώ από αυτά τα χρήματα. Επισκεφτείτε την περιοχή και κάνετε τη δική σας αξιολόγηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Έχετε κάθε δικαίωμα να εκφράζετε τις εντυπώσεις σας, αλλά εγώ ω επίτροπο θυμάμαι ότι εμεί ήμασταν εδώ, μιλήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιλήσαμε στου βουλευτέ. Είχατε έρθει στο γραφείο μου και όχι μόνο ο Τζέρι Άνταμ, αλλά και άλλοι βουλευτέ. Και θυμάμαι και τι ε, επισκέψει, όχι μόνο στο Μπέλφαστ που έκανα εγώ. Εγώ πήγα σε, ε, στην σε διάφορα σημεία, μίλησα με νέου ανθρώπου οι οποίοι δούλευαν για την ειρήνη σε επίπεδο δρόμου. Και συνεργαστήκαμε. Πιστεύω ότι η διαδικασία λειτουργήσε από τη βάση πώ τα πάνω. Ήταν μια εξαιρετικά αποτελεσματική συνεργασία. Ε, βέβαια, συμφωνώ μαζί σα όταν λέτε ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Και ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει τον ενδιαφέρον τη ακόμη πιο έμπρακτα. Σύμφωνοι. Ελπίζω ότι κάποια μέρα θα επιστρέψουμε ω ε, Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων για να δούμε πραγματικά τι άλλαξε και τι άλλο μένει να κάνουμε. Πατ ε, αλλά η είναι, είναι εδώ. Είναι από την Επιτροπή Γεωργία και ζήτησε τον λόγο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πλέον εδώ. Και ο είναι ο ο ομιλητής. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λίντεμανς ε, για την επισκόπηση και για την ενημέρωση για την κατάσταση όχι μόνο για τη διαδικασία συμφελήσεως αλλά και για το Διεθνέ Ταμείο για την Ιρλανδία το οποίο συστήθηκε το 1995 και το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία και δημιούργησε 55.000 θέσει εργασία, κάποια προγράμματα, 130 από την Ευρώπη και φυσικά ε, όλα Αυτά ε, ήταν το αρχικό κεφάλαιο που κατέληξε και σε πρόσθετη χρηματοδότηση από άλλες πηγές. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά στο Κοινοβουλίο όταν ε, ε, ξεκίνησε η κατάπαυση πυρός τότε ο Ζακ Ντελόρ απάντησε και είπε ότι η Ευρώπη θα απαντήσει με ένα θετικό και πρακτικό τρόπο και η μόνη δομή που υπήρχε τότε ήταν να αυξηθούν οι εισφορές με το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία ε, τότε διασφαλίστηκε και από τον Αρμόδιο Επίτροπο ότι θα χορηγούνταν πρόσθετοι πόροι και φυσικά αυτό μας οδήγησε στην ειρήνη και στη συμφιλίωση και ε, είχαμε ε, την έναρξη της διαδικασίας στο Belfast ε, και νομίζω ότι οι τρεις ε, βουλευτές, ευρωβουλευτές από την Βορειοελλανδία ήταν εκεί και ο Ιεν και ήταν, συμμετείχαν στη διαδικασία εκείνη τη στιγμή, είχαν τεθεί κάποιοι στόχοι και συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τους στόχους αυτούς, ε, αλλά ε, και οι δύο πλευρές ε, συνεργάστηκαν. Εγώ εκπρόσωπούσα πέντε από τις έξι επαρχίες και ε, μπορώ να σας πω ότι είχαμε και πέντε μίλια ε, σύνορα από ε, το βορρά. Εγώ όταν μεγαλώνω πίστευα ότι δεν ήταν η πρωτεύουσα γιατί ήταν πιο κοντά σε εμά και αντί να έχουμε την... και δεν είχαμε πολλές φορές την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Δουβλίνο. Το Δουβλίνο. Έτσι λοιπόν ε, είχε συμφωνηθεί ότι ε, θα υπήρχε χρηματοδότηση και από τα δύο ε, ταμεία για αυτές τις επαρχίες ε, που βρίσκονταν στην Περμεθόριο γιατί εκεί τα προβλήματα μπορεί να μην ήταν τόσο ανθρωπιστικά αλλά ήταν κυρίως εμπορικά. Όμως ε, ωφελήθηκαν πάρα πολύ λόγω του IFI, του Διεθνούς Ταμείου την και από τη διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης. Ε, ίσως δεν ήταν όλες οι πρωτοβουλίες από τη βάση, αλλά ήταν σε μεγάλο βαθμό. Και εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές των κινητήτων και από τις δύο πλευρές των συνόρων συνεργάστηκαν και αυτό γίνεται χάρη στα διάφορα προγράμματα που συμπεριλαμβανόταν ε, στο πρόγραμμα PIS και χάρη στο IFI. Και χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα την Κομισιόν να λέει ότι υπάρχει μια δυνατότητα. Εγώ ποτέ δεν συμφώνησα με την απόφαση που ληφθήκε ότι το Διεθνέ Ταμείο για την Ιρλανδία θα πρέπει να σταματήσει ε, τη χρηματοδότηση το 2010 ε, και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι υπάρχει δυνατότητα ε, και η Κομισιόν θα σκεφτεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες του Ταμείου μπορεί να είναι περιορισμένες και μπορεί να γίνει εστίαση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτό φυσικά ανάλογα και με τις δημοσιονομικές προεπτικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά ξεκολουθώ να πιστεύω ότι από την πρόσθετη χρηματοδότηση μπορούν να προκύψουν ωφέλη που θα πολλαπλασιάσουν τα ωφέλη του ΠΙΣ 4 και ξέρω ότι ε, ε, και ε, οι κατοικοί θέλουν να μιλήσουν ε, με τους, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά κυρίως με τον Τζιμ Μάικλσον, την Μπάρμπαρα Λεμπρούν και τον Τζον Μάικλσον που είναι βουλευτές από τη Βόρεια Ιρλανδία και Φυσικά οι πολιτικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο συνεργάζονται και αυτό ανεξάρτητα από ε, ποιο ρεύμα εκπροσωπούν. Όλοι οι επικεφαλείς των κομμάτων συνεργάζονται και εργάζονται και στο Μπελφέστ και στο Δουβλίνο και στο Λονδίνο. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος ε, ε, δωρητής για το IFI και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να συστήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για την περίοδο 2010-2013 και ελπίζω και, η Ευρωπαϊκή, και οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία να συνεισφέρουν επίσης για να μπορέσουν να επιτρέψουν ε, στο Ταμείο να συνεχίσει τη λειτουργία του. Το PIS 4 είναι απολύτω απαραίτητο και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με όσου δραστηριοποιούνται και επιτόπου, αλλά και μεταξύ μα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φυσικά είναι αλήθεια ότι ενώ προγράμματα ε, ξεκινούν, κάποιος μπορεί να είχε την εντύπωση ότι ήταν ε, μόνο υπό την ευθύνη του Δουβλίνου και του Λονδίνου. Είναι πολύ σημαντικό και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνο απαραίτητο ε, γιατί εμείς ως άτομα θέλουμε να ε, δοξαστούμε λόγω αυτής της διαδικασίας, αλλά θέλουμε να τονίσουμε και πώς διαδραματίζει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, θέλω να αποτίσω φορό τιμή σε εσά και για το χρόνο που αφιερώσατε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά είμαι σίγουρος ε, και ε, ο σημερινός Επίτροπος αλλά και ο επόμενος Επίτροπος θα συνεχίσει το καλό έργο. Ο ΣΕΜ και πάλι. Πολύ σύντομα. Δεν διαφωνώ με τον συνάδελφο Νίκολσον, απλά όταν αναφέρα κάποια ονόματα ήθελα να τονίσω ότι για εσύ και από τις δύο πλευρές ε, εκείνη ε, την περίοδο ε, ε, υπήρξε και νομίζω ότι και ο Τζακ Νίκολσον ανέλαβε ηγετικό ρόλο και φυσικά και ο Ζακ Ντελόρ και αυτό ουσιαστικά καταδεικνύει αυτό που λέω ότι δεν αναγνωρίζεται ο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαρκώς για όσα έχει κάνει και άκουσα τι είπε και ο Τζιμ και για το Βορράλ και για τον Νότο. Αν ρωτήσετε του περισσότερους ε, για το AFI θα σα πούν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Και επίση, ε, συμφωνώ πολύ με τον Τζιμ και με τον Πατ ότι οι Ευρωβουλευτέ θα πρέπει να εμπλέκονται πολύ περισσότερο σε όλα. Είναι το δημόσιο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν ε, δεν συμμετέχουν τότε ε, δεν ε, εντυπώνεται στο μυαλό των ανθρώπων η Ευρωπαϊκή Ένωση και για οποιαδήποτε προγράμματα ξεκινούν θα πρέπει να εμπλεκόμαστε περισσότερο. Και φυσικά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαδραματίσαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία καθ' όλη τη ε, διάρκεια της διαδικασίας αυτής και η δράση τους θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Ευχαριστώ. Να ξαναδώσουμε το λόγο στην κυρία Λίντεσμαν για να απαντήσει στα σχόλια που ακούστηκαν. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, για το ενδιαφέρον που δείχνουν για τη δράση της Κομισιόν, ε, για το ΠΙΣ και για το ΑΕΦΑΙ για τις διάφορες παρατηρήσεις ε, που ακούστηκαν καταρχήν για την έλλειψη δημοσιότητας. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε κάποιες δυσκολίες στο να διαδίδουμε τις επιτυχίες μας, ε, τις, όσα κάνουμε στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΙΣ στο πλαίσιο του προγράμματος συνοχής, αλλά και με το IFI. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σε επίπεδο Επιτροπής Κομισιών είναι ότι κατά τη διάρκεια των ε, ανοιχτών ε, ημεριδών που οργανώνουμε μαζί με την Επιτροπή, με την ΚΑΜΑ είναι να παρουσιάσουμε και κάποια εργαστήρια ε, και προσπαθούμε να απευθυνθούμε και σε ένα ευρύτερο κοινό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τους παρουσιάσουμε ποια προσέγγιση έχουμε ακολουθήσει μέσω του προγράμματος PIS και να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούν να διαδοθούν οι βέλτιστες και οι καλές πρακτικές σε παρόμοιες καταστάσεις. Παραδείγματο χάρη, φέτο το εργαστήριο έγινε ε, με δύο παρουσιάσει που είχαμε από δύο διαφορετικέ πόλει, Μάλμο και Ρότερνταμ, και οι παρουσιάσεις αυτές αφορούσαν και το πώς διάφορες προσεγγίσεις μπορούν να βοηθήσουν τις κοινότητες να κατανοήσουν καλύτερα η μία την άλλη, να συνεργαστούν και να ζήσουν καλύτερα μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε ποια είναι τα θετικά και να παρουσιάσουμε σε όλους τους ενδιαφερομένους ε, τι έχουμε κάνει με το πρόγραμμα PIS και ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές, ποια είναι τα διδάγματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, ανοιχτές ημέρες είχαμε ένα πάνελ όπου ε, δύο επίτροποι, Βασίλη και Φένο, ε, παρουσίασαν πώς μπορούμε να φέρουμε κοντά παιδιά από διάφορες κοινότητες και πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε την ειρήνη σε τέτοιες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε πραγματικά να διαδώσουμε τι πράττουμε, αλλά και άλλα πρέπει να γίνουν, κυρίως όταν αναφερόμαστε ε, στην Ιρλανδία όταν ε, ρωτά κανείς για τον IFI πράγματι οι πολίτες σκεφτούνται περισσότερο την πρωτοβουλία των ΗΠΑ και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς ε, θέλαμε να διασφαλίσουμε με το IFI ότι και είναι ορατή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε μέσω του IFI σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο έργο που κάνουμε μέσω του PIS και του AFI. Ξέρω ότι δεν ε, ήρθαν σε επαφή με τον κύριο Μπαρόσο οι ευρωβουλευτέ κατά την επισκευσή του στην Βόρεια Ιρλανδία. Ήταν ε, μια απόφαση που λήφθη την τελευταία στιγμή ε, από τον κύριο Μπαρόσο να προσγειωθεί στην Ιρλανδία γιατί νομίζω επέστρεφε από τι ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν ήταν απόφαση τελευταία στιγμή κατά κάποιο τρόπο και ήταν δύσκολο να οργανωθεί σωστά η επίσκεψη. Αλλά λαχθέντως αυτό το σημειώνω αυτό που είπατε και θα επενδυθώ στον πρόεδρο της Tax Force ε, της Βόρειας Ιρλανδίας και θα δω μαζί του σε ποιο βαθμό μπορούμε να μπλέξουμε και καλύτερα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην, ε, στις εργασίες της Task Force. Σημείωσα και τα προβλήματα εφαρμογή που αναφέρετε, τη γραφειοκρατία που ενέχεται για την παράδοση αποτελεσμάτων ε, από το πρόγραμμα PIS. Εμεί θεωρούμε ότι καλά τα πάει το πρόγραμμα. Ε, έχουμε πετύχει τους στόχους ό,τι αφορά τις αναλήψεις ε, υποχρεώσεων ε, αν και καταλαβαίνουμε ότι τα ίδια αυτά των προγραμμάτων δεν είναι εύκολα μικράμε για πολύ μικρά σχέδια και χρειάζεται χρόνος να συσταθούν και για να έχουμε αποτελέσματα αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με το πώς προοδεύουν τα πράγματα αλλά φυσικά θα απευθυνθούμε στην διαχειριστική αρχή και θα δούμε αν έχει συγκεκριμένε ανησυχίε σε σχέση με την εφαρμογή, την γραφειοκρατία ή σε σχέση με διαδικασίε που είναι δύσκολο να συνεχιστούν στο πλαίσιο του προγράμματο ΠΙΣ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι διάφορε επεμβάσει για το μέλλον των δύο μέσων οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα σε κάπως διαφορετικό πλαίσιο. Όταν καταρχήν ε, εξετάσουμε το IFI, ε, μέχρι φέτος είχε προβλεφθεί συνεισφορά από τον κοινοτικό προπολογισμό και τώρα εξετάζουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσθετη συνεισφορά στο Ταμείο στο πλαίσιο των σημερινών διανομιστικών προοπτικών για το 2011, 2012 και 2013 δηλαδή το ανανεωμένο ενδιαφέρον για να συνεχιστεί συνεισφορά στο ΕΕΦΑ e πυροδοτήθηκε από ένα ενδιαφέρον ε, των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεχίσουμε με το μέσο. Η απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, λόγω των εκλογών εκεί. Ε, υπάρχει η εξέταση του ζητήματος, όμως αυτό ήταν το στοιχείο που έκανε το, τις δύο χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, να προσεγγίσουν την Κομισιόν και να δούμε και σε ποιο βαθμό από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να υπάρξει μια δέσμευση για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ταμείου. Το θέμα είναι ότι αφενός ε, πρέπει στα πλαίσια των σημερινών δημοσιονομικών προοπτικών να βρούμε διαθέσιμους πόρους και Επίσης πρέπει να συστήσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και εδώ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν να αποφασιστεί η συνέχιση του Ταμείου. Τώρα για το πρόγραμμα PIS διαφέρει κάπως το πλαίσιο, είναι πιο απομακρυσμένο στον βαθμό που το PIS 3 θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος αυτών των δημοσιονομικών προοπτικών, μέχρι τα τέλη του 2013 δηλαδή. Και έτσι λοιπόν η συνέχιση του PIS θα πρέπει να αποφασιστεί στο πλαίσιο των συνολικών αποφάσεων που θα ληφθούν για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Δηλαδή το ποσό που θα αφιερώσουμε στην πολιτική συνοχή και να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα για ένα ps 4 στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού φακέλου για την πολιτική συνοχή. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, για την ε, περιφερεια... όταν ε, συζητήσουμε για την εδαφική συνεργασία μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε την κυρία Λίντερμαν. Ο κύριο Νίκολσον θέλει να πει κάτι. Ναι, πολύ σύντομα χαιρετίζω αυτά που είπε η κυρία Λίντερμαν. Όμω πρέπει να πω ότι στην ουσία δεν σας είπα σήμερα εδώ κάτι που δεν είδα επιτόπου. Και έχετε δίκιο κυρία Πρόεδρε. Ε, είναι σημαντικό να επισκεπτόμαστε τα διάφορα project και να βλέπουμε τι γίνεται. Αν όμως αμφιβάλλετε για αυτά που λέω, μην πάτε εκεί που ε, το EDFS ή το SUPP σας είπαν να πάτε στο Belfast και στην Ιρλανδία. Πηγαίνετε να μιλήσετε με τις ε, οργανώσεις ε, και τους ανθρώπους που έχουν μεγάλες δυσκολίες να βρουν υποστήριξη. Αυτά που σας λέω σήμερα στην ουσία είναι ότι υπάρχει ε, ε, μεγάλη ανάγκη να δώσουμε μεσοπρόθεσμα ε, μία αξιολόγηση σχετικά με το πώς θα πάει η Task Force. Αυτή η ενδιάμεση επισκόπηση είναι κάτι που χρειαζόμαστε και φυσικά δεν θα ζητήσω από τα να μου πει αν το, χρειαζόν, το χρειάζονται ή όχι. Θα μας πούνε ότι δεν το χρειάζονται. Εγώ θα δω αν λειτουργεί το πράγμα ή όχι. Αυτό ζητώ λοιπόν από σας σήμερα και χαίρομαι να παίζω κάποιο ρόλο. Δεν θέλω ε, να εμπλέξω περισσότερους βουλευτές ή όχι. Όταν οι άνθρωποι της ε, Βόρειας ε, Ιρλανδίας σκέφτονται την Ευρώπη, σκέφτονται τους ευρωβουλευτές. Σε αυτούς μιλάνε, σε αυτούς απευθύνονται. Γι' αυτό σας μιλάω σήμερα και σας ζητώ να πάτε στην Κομισιόν και να ζητήσετε μια ενδιάμεση επισκόπηση, να δουν ποια είναι τα λάθη. Δεν υπάρχει αρχή σε, αυτή, σε αυτόν τον κόσμο που να μην κάνει λάθη. Να βρούμε ποια είναι τα λάθη, να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε και να συνεργαστούμε σε αυτό. Ευχαριστούμε, James. Θα σημειώσουμε το σχόλιο σου, θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη, θα επανέλθουμε ε, στην Κομισιόν να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Κλείνω. Η συνεδρίασή μας ακυρώνεται το σημείο 9 λόγω απουσίας ε, της κυρίας Καρόνσα και θα επανέλθουμε στις 3. Και να δούμε και ποιοι είναι οι συνάδελφοι που δεν μπόρεσαν να έρθουν στις Βρυξέλλες ακόμα, να δούμε πώς θα γίνει με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ.